Καλησπέρα. Ξεκινάμε. Να σας ενημερώσω ότι η συνάντηση ακούγεται και μεταδίδεται από το ίντερνετ. Σας ενημερώνω όπως οφείλει. Έχετε λάβει στις 10 Δεκεμβρίου το σχέδιο ημερησίας διάταξης. Στο πρώτο τμήμα της συναντησής μας σήμερα το απόγευμα θα ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο κ. Σεύκοβιτς που ανήγγειλε ότι θα έρθει σε κανένα πεντάλεπτο. Μπορούμε να σα κάνουμε κάποιες άλλες ενημερώσεις στο μεταξύ. Ο κ. Τσεύκοβιτς θα μας ενημερώσει για τον κανονισμό σχετικά με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και θα μας δώσει τις απόψεις του για την έκθεση Γκουρμάη σχετικά με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Κατόπιν θα έχουμε μια δεύτερη ακρόαση στις 4.30 το απόγευμα. Θα μιλήσουμε με τους αντιπρόεδρους κύριο Μικελάνχελ Μαρτίνες και κύριο Ότμαρ που είναι υπεύθυνοι για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και που θα μας μιλήσουν για τις δύο τελευταίες συναντήσεις της ΚΟΖΑΚ, αυτή που έγινε στο Δουβλίνο το πρώτο εξάμεινο και αυτή που έγινε στο Βίλμιους για το δεύτερο εξάμεινο όπου είχαμε, δεν μπόρεσα να μετάσχω και εγώ διότι όπως ξέρετε είχαμε στείλει μια αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον άρα θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και για μέ να, να ξέρω τις πληροφορίες που προέρχονται από την δεύτερη αυτή ιδίω συνάντηση της ΚΟΖΑ. Κάπου το απόγευμα θα έχουμε τον τριμερή διάλογο με, για τα πολιτικά κόμματα. Αύριο θα ξεκινήσουμε στις 10, όπως ζητήσατε εσείς, αποφασίσαμε η συνάντηση των συντονιστών να γίνει 9, αύριο, και όχι σήμερα μετά τη συνεδρίαση. Άρα 9 με 10 θα έχουμε συνάντηση συντονιστών και κατόπιν μετά τις 10 κανονική συνεδρίαση όπου θα ψηφίσουμε την έκθεση David Martin για την Εξεταστική Επιτροπή. Έχει αναγγελθεί αυτό εδώ και καιρό πρέπει να κλείσουμε. Κατόπιν θα ακούσουμε την έκθεση του Αντιπρόεδρου κ. Μόρτεν Μέσορ Σμιτ για την αλλαγή των άθρων 166 και 195 του κανονισμού και τέλος έχουμε το σχέδιο έκθεσης για Τερμέκη για την διαδικασία ανάκλησης και προάσπισης της κοινοβουλευτικής ασυλίας. Αύριο επίσης θα συζητήσουμε την έκθεση Ράνζελ για την ενεργοποίηση της συνθήκης, για την υλοποίηση της συνθήκης της ε, Λισαβόνας και αν το επιτρέψουν οι συντονιστές αύριο το πρωί και συμφωνήσουν θα έχουμε και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το περιεχόμενο της γνωμοδότησής μας σχετικά με την έκθεση της έκον για τις δραστηριότητες της Τρόικα. Αν δεν έχουμε αντιρρήσει, θεωρώ ότι εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη. Έτσι είναι. Πάμε στο δεύτερο σημείο. Μία ενημέρωση του κειμένου που έχουν υποβάλει οι ερευνητικέ υπηρεσίες ε, μελετών για το τις διαδικασίες επικύρωσης που συνεχίζονται αυτές σε κάποια κράτη, ιδίω για τις ε, συνθήκες σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Σημείο 3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη συνεδρίαση τη 24 Οκτωβρίου του περασμένου έτους είναι διαθέσιμο και θα εγκριθεί αν δεν υπάρξουν ενστάσεις από πλευρά σας. Φτάσαμε κατόπιν στο σημείο 4, χωρίς ωστόσο τον κύριο Σεύκοβιτς. Ή διακόπτουμε ή προχωράμε. Ε, λοιπόν, δεν έχουμε το 7. Λοιπόν, διάλειμμα, σύντομη διακοπή μέχρι την άφηξη του κύριου Σεύκοβιτς που έχει κολλήσει στην κυκλοφορία. Θα φτάσει σε πέντε λεπτά. Allora, possiamo riprendere i nostri lavori. Μπορούμε λοιπόν να επαναλάβουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας, καθότι ήλθε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Εύκοβιτς. Υπό το σημείο 4 λοιπόν της Μερίσιας Διάταξης θα συζητήσουμε την πρωτοβουλία των πολιτών, ένα ζήτημα το οποίο ενεγράφει στη Μερίσια Διάταξη κατόπιν δικού σας αιτήματο μετά τη συνάντηση της 4 η Σεπτεμβρίου και μετά την αξιολόγηση της κατεξουσιοδότηση πράξης της Κομισιόν. Μπορούμε να τη βελτιώσουμε όμως ακόμη περισσότερο αυτή την αξιολόγηση της ε, πρωτοβουλίας, αν θέλουμε να βελτιώσουμε και την ίδια την πρωτοβουλία. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να έχουμε αυτό το διάλογο με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς, για να δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να βελτιώσουμε την όλη διαδικασία ακόμη περισσότερο. Είχα ζητήσει ε, από τον Υπουργό Εξωτερικών να έλθει, αλλά δεν ε, μπόρεσε, είχε αγγελμένες υποχρεώσει. Έχουμε όμως ε, τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Σεύκοβιτς, με τον οποίο θα δείξουμε και άλλα θέματα που ξέρω ότι απασχολούν συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προφορική μάλλον έκθεση γκουρμάι, να καλυφθούν ε, και οι γραπτές ερωτήσεις. Ή μήπω να μιλήσει πρώτα κύριε Γκουρμάη και να δώσω μετά το λόγο στον κύριο Σεύκο για να μα τα πει. Όχι. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Σεύκοβιτς. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να συζητήσουμε τα πολύ σημαντικά αυτά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, όπως προτείνατε και εσείς, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρωτοβουλία των πολιτών. Όπως γνωρίζετε, τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου του 2012 παρά μια διστακτική αφετηρία, το συζητήσαμε επανειλημμένως. Τώρα νομίζω ότι αυτό το διακρατικό εργαλείο της άμεσης δημοκρατίας ε, έχει πάρει πλέον ε, ε, έχει μπει στην κανονική του τροχιά και λειτουργεί τουλάχιστον 21 πρωτοβουλίες έχουμε καταγράφει μέχρι τώρα 10 εκ των οποίων για 10 από τις οποίες έληξε η περίοδος συλλογής δύο αποσύρθηκαν από τους οργανωτές. 9, προτινόμενες πρωτοβουλίε συνεχίζονται ακόμη. Είναι σε εξέλιξη και καλύπτουν διάφορα θέματα, το περιβάλλον, την παιδεία, τι τηλεπικοινωνίε, τα μίντια, τα δικαιώματα των πολιτών, τα δικαιώματα των καταναλωτών και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι καλύπτονται ζητήματα ε, που ενδιαφέρουν πάρα πολύ ε, του πολίτε, είναι κοντά στο μυαλό και την καρδιά του. θα έλεγα και είναι ενθαρρυντικό ο αριθμό των πρωτοβουλειών, δείχνει τον ενθουσιασμό των πολιτών και τη δέσμευσή του ε, σε αυτό το νέο δικαίωμα. Επιπλέον, τρεις από τις δέκα ε, ήδη διεκπαιρεωθήσεις πρωτοβουλίες για κάποιες έχουν ε, συλλεγεί οι απαιτούμενες υπογραφές. Πρέπει βέβαια να παληθέσουμε τον αριθμό της υποστήριξης αυτής, αλλά νομίζω ότι υπόσχεται πολλά για το μέλλον ε, του δημοκρατικού μέσου η όλη αυτή διαδικασία. Εξακολουθούμε βέβαια να μαθαίνουμε και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την πρωτοβουλία των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Διότι πιστεύω ότι είναι και αναπόφευκτο αυτό λόγω της κλίμακας του καινοτόμου χαρακτήρα αυτής της πρωτοβουλίας. Για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο σε τόσο ευρία κλίμακα, σε επίπεδο δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι συνολικά αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν συλλέξει πάνω από πέντε ε, εκατομμύρια υπογραφές, 5 εκατομμύρια πολίτες δηλαδή έχουν ήδη συμμετέχει και υποστηρίξει μια από αυτέ τις πρωτοβουλίες και νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το νούμερο αυτό. Πόσοι Ευρωπαίοι πολίτες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο δημοκρατικό του δικαίωμα με την πρώτη δυνατή ευκαιρία και πιστεύω ότι θα το συνηθίσουν και θα το χρησιμοποιούν ε, αυτό το δικαίωμα ακόμη περισσότερο και πιο συχνά στο μέλλον. Ιδίω όταν βλέπουν ε, να αφορά ένα θέμα που τους ενδιαφέρει πολύ και θα θέλουν τότε να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα σημαντικά ζητήματα που είναι στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι ως Κομισιόν για το ότι θα μπορούν οι πολίτες να αξιοποιούν πλήρως αυτό τους το νέο δικαίωμα και στην ιστοσελίδα της Κομισιόν και στο Μητρό. Είδαμε ότι αυτά τα δύο ε, είναι ένα ισχυρό εργαλείο και προσπαθούμε να τα προσπαρμόσουμε και τα δύο και στις απαιτήσει και στις νέες εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει μετά τη θέση αρμογευτή οδηγία. της ε, Και βέβαια αυτή η οδηγία δεν είναι μόνο μια πηγή πληροφοριών για τις πληροφορίες, έτοιμα καταχώρησης, για παράδειγμα, ή κάποιες, κάποια έτοιματα που απορρίφθηκαν, αλλά είναι και μια διαπαφή, ένα interface μεταξύ της Κομισιόν και των οργανωτών και τους επιτρέπει επίσης ε, πιο εύκολα να προσθέτουν καλύπτουν ε, άλλες γλωσσικές εκδοχές, ε, να προσαρμόζονται τη χρηματοδότηση και να ε, απευθύνονται στην Κομισιό και στις υπηρεσίες της για κάποιες ερωτήσεις. Είναι ένα είδος φόρουμ όπου οι διάφορες υπηρεσίες και οι οργανωτές συνεργάζονται και ήταν πολύ αποτελεσματικό. Τώρα το λογισμικό της Κομισιόν διατίθεται δωρεάν. Το χρησιμοποίησαν όλες οι πρωτοβουλίες, δηλαδή όσοι συνέλεγαν online τις υπογραφές το επικαιροποιούμε και το βελτιώνουμε συνεχώς το λογισμικό αυτό, διότι στον τομέα αυτό έχουμε βέβαια συνεχώς ε, καινοτομία με την ε, ψηλότητα ταχύτητα και χρειάστηκε να κάνουμε τις απαραίτητες δοκιμές ε, και στις μοναδιές αντοχής, λειτουργικότητας ευαλωτότητας, διότι φυσικά όταν μιλάμε για ένα εκατομμύριο προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτό το εργαλείο, ώστε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να τηρείται, να γίνεται σεβαστή και να προστατεύονται τα δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα. Ε, αντιμετωπίσαμε κάποιες αρχικές δυσκολίες, ε, σε επίπεδο δηλαδή οργανωτών δεν ήταν εύκολο να βρουν έναν προσιτό πάροχο εμείς ξεπεράσαμε την υποχρέωσή μας ε, δυνάμει του κανονισμού και ξέρετε ότι ως προσωρινή ε, προαιρετική λύση ε, τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιούν δωρεάν τους διακομιστές που έχουμε στο Λουξεμβούργο. Υπήρχε μέχρι την 1η Νοεμβρίου η προθεσμία και την ξεπεράσαμε ε, επειδή είχαμε, όπως σας είπα, μια διστακτική αρχή, θέλαμε να πελκιστοποιήσουμε ε, την κατάσταση, την ασφάλεια του λογισμικού και οι οργανωτικές επιτροπές αντιμετώπισαν προβλήματα με την παράδοση υπό της προθεσμίας και με την ανάληψη οικονομικών ε, για την κατάσταση του λογισμικού και την ε, ασφάλειά του. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την συλλογή υπογραφών για τις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ένα άλλο θέμα για το οποίο χρειάστηκε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη ήταν ο εξαρθολογισμός της διαδικασίας που σχετίζεται με την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης, statements of support. Αυτό θυμάστε ότι ήταν και ένα από τα δυσκολότερα κομμάτια τη διαπραγμάτευση. Είναι και μακροσκελέο στο παράρτημα για αυτόν τον λόγο. Επειδή σε κάθε κράτο μέλο οι απαιτήσει ήταν λίγο διαφορετικέ για τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονταν προκειμένου να προχωρήσουν με την επαλήθευση εγκαίρω και ομαλά. Η συζήτηση έγινε με τα κράτη-μέλη σε επίπεδο ομάδας εργασίας, με πυρογνώμονες από τις ε, αρμόδιες αρχές και επικεντρώθηκε στα δύο σκέλη διαδικασία, διαδικασίας, ε, το, την πιστοποίηση, το σύστημα πιστοποίησης ε, και αυτές τις δηλώσεις υποστήριξης. Και το θέμα της απλώστευσης των δεδομένων που θα πρέπει να παρέχουν οι υπογράφοντες εξετάστηκε σε αυτή την ομάδα εργασίας, και τον Ιούλιο ως αποτέλεσμα εγκρίναμε με της πράξη τροποποίηση ε, των απαιτούμενων δεδομένων για έξι κράτη-μέλη. Σε περισσότερες περιπτώσεις ε, η απλουστευμένη διαδικασία οδήγησε σε μείωση του αριθμού των πολιτών που στερούνταν του δικαιώματο αυτού λόγω της παρέκκλησης, λόγω, των ε, αντιφάσεων σε αυτά τι απαιτήσει για τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης δίθηκε πρώτη φορά πιστοποίηση για κάποια αιτήματα. Ομαλή διαδικασία μέχρι τώρα. Και οι οργανωτές θα μας παρουσιάσουν επαληθευμένες υπογραφές, πιστοποιημένες υπογραφές, ίσως και πριν από τα Χριστούγεννα. Αν η επαλήθευση είναι θετική, τότε μετά θα αναλύσουμε κάθε μία από τις πρωτοβουλίες αυτές. Νομικός, ξέρετε, ότι δεν υποχρεούμαστε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της πρωτοβουλίας, αλλά πάντοτε θα δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή, θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλη σοβαρότητα της ε, πρωτοβουλίας και μετά θα αποφασίσουμε αν θα αναλάβουμε δράση ή όχι. Θα θυμάστε και από τις διαπραγματεύσεις, η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει διαδικασια εξέταση, περιλαμβανει ακρόαση που θα ε, πρέπει να διοργανώνεται εδώ στο Κοινοβούλιο με εκπροσώπηση της Κομισιόν. Αυτό το προβλέπει ο κανονισμός και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε οι οργανωτές να μπορούν να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους αναλυτικά και άλλοι ε, ενδιαφερόμενοι να μπορούν επίσης να εκφράζουν τις απόψεις τους. Και αυτό θα μπορεί να γίνει μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Κομισιόν, για να μπορεί ε, στην ανακοίνωση που θα πρέπει να εγκρίνει η Κομισιόν ε, να μπει και το πόρισμα αυτής της δημόσιας ακρόασης. Έχω και ένα έτοιμο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό η right to water να μας στήσει να δεχθούμε τους ε, επαληθευμένους, ε, τους πιστοποιημένους αυτούς ε, υπογράφοντες. Και μετά θα πρέπει να βασιστούμε και σε όλη αυτή τη δικασία για να εκδώσουμε την ανακοίνωσή μας για αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών. Θα μπορούσε λοιπόν ε, για την ε, οργάνωση Riot του Water και τη σχετική πρωτοβουλία δικαιώματο στο νερό να ε, οργανωθεί γρήγορα μία δημοσία κρόαση από το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα της συζήτησης. Το Μάρτιο το αργότερο θα πρέπει να έχουμε εκδώσει αυτήν την ανακοίνωση με την προθεσμία των τριών μηνών. Είμαστε σε επαφή και με την Οργανωτική Επιτροπή Right to Water για να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση ψηλού επίπεδου μεταξύ των οργανωτών και των αρμόδιων επιτρόπων και υπηρεσιών της Κομισιόν. Και πιστεύουμε ότι και η δημοσιακρόση και η συνάντηση των Κομισιόν θα μπορούσε να είναι λίγο πολύ στην ίδια ημερομηνία για να είναι πιο εύκολο για τους οργανωτές. μέσα σε μια μέρα δηλαδή να παραστούν οι εκπρόσωποι της Οργανωτικής Επιτροπής και στις δύο αυτές συναντήσεις. Αν μπορείτε λοιπόν τον Ιανουάριο να οργανώσετε αυτή την δημόσια κράση θα σας ήμουν ευγνώμος. Ολοκληρώνοντας θα σας πω, το 2013 τότε των Ευρωπαίων Πολιτών, χάρη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αυτό το νέο δημοκρατικό εργαλείο ε, το καταστήσαμε πολύ πιο γνωστό Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη από ό,τι προηγουμένω. Όλε τι εκδηλώσει που αφορούσαν το έτο των πολιτών τι αξιοποιήσαμε για να προβάλλουμε αυτό το νέο δικαίωμα του πολίτη. Για να νιώθει ο πολίτη ε, ότι του ανήκει όλη αυτή η διαδικασία και μέσω αυτή τη συμμετοχική άμεση επικοινωνία μεταξύ με το Κοινοβούλιο, με του ευρωπαϊκού θεσμού εν γέννη, θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχιστεί αυτό. Και να ενθαρρύνουν οι πολίτες, ή μάλλον ε, τα κράτη-μέλη, αλλά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους πολίτες να ασχολούνται ε, με την πρωτοβουλία αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και σημαντικό και για τις προσεχείς ευρωεκλογές για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Σταματώ εδώ, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να παρακολουθήσω τη συζήτηση, αν χρειαστεί να απαντήσω σε ερωτήσει και μετά, όπω είπατε, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ε, ε, ευχαριστώ. Η κυρία Γκουρμάη ζήτησε καταρχά το λόγο. Καταρχήν, ως ε, συνεισηγήτρια. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το τι πιστεύουν τα δύο μέρη για το σημαντικό αυτό μέσον που δίνει ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες να ε, ε, εκφράσουν τις απόψεις τους και να θυμηθούμε ότι εδώ είναι χαρτογράφητα νερά, δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό θέλαμε επανεξέταση στα τρία χρόνια για να είμαστε βέβαιοι ότι αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά θα διορθωθεί. Ένα χρόνο είχε πει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σεύκοβιτς. Είναι σημαντικό να ακολουθηθεί λοιπόν σωστή διαδικασία. Πολύ σημαντικό είναι ότι χειρίζεστε με την καταπληκτική σας ομάδα το χαρτοφυλάκιο αυτό και πρέπει εδώ να τους ευχαριστήσουμε για όλη αυτή τη δουλειά και σας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανταλλαγή απόψεων σε ε, ε, περιόδους κέρυες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Επίτροπος ε, ε, είχε μιλήσει και για ευρωπαϊκή ηθαγένεια και όχι μόνο ευρωπαίους πολίτες. Ο Αλέν Λαμασούρο, ο μεγάλος συνεισηγητής μου, δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Και εκείνο όμως πιστεύει ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε καλή δουλειά συμφωνούμε ότι οι βασικές προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν στο μέλλον, γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Ο αριθμός των πρωτοβουλειών που υποβλήθηκαν μέχρι τώρα ε, με κάνουν αισιόδοξη, γιατί είναι, αντικατοπτρίζουν καινούργιες ιδέες και πρέπει να μελετήσουμε τι υπάρχει. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες άρχισαν να βλέπουν την προστιθέμενη αξία από όλα αυτά. Δεν γίνονται όλα εν μια νυχτή, είναι μια διαδικασία εξελικτική, αλλά η θετική εξέλιξη δεν κρύβει τις τεχνικές δυσκολίες που είχαν οι διοργανωτές ε, μέχρι τώρα και ακόμα υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις. Όταν ε, καταρτίζαμε τον κανονισμό ε, γνωρίζαμε ότι δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα αφού ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτή η πρωτοβουλία σε τόσο μεγάλη κλίμακα με τον Αλέν Λαμασούρ κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν, ούτω ώστε αυτό το εργαλείο να είναι φιλικό προς το χρήστη και τον πολίτη. Ούτως ώστε να υπάρχουν και να... γιατί υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες. Η δυσκολία για τους διοργανωτές ήταν τεχνικής φύσεων και αυτό είναι καλό. Γιατί ε, αν είναι τεχνικής φύσεως οι δυσκολίες μπορούμε να τις διορθώσουμε και το πρόβλημα του online server για τη συλλογή υπογραφών ελήθηκε εν μέρη με τη βοήθεια της Κομισιόν, είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, αλλά πρέπει να βρούμε και κατάλληλη λύση και θέλω να ακούσω τι λέτε κι εσείς εδώ. Γιατί υπάρχουν σχετικά αιτήματα και περιμένουν και κατάλληλες απαντήσεις οι πολίτες. Να τους πούμε δηλαδή, ε, κάντε υπομονή και θα δώσουμε λύση μέχρι τότε. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα στα πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού. Πρέπει να φροντίσουμε να απαλείψουμε όλα τα εμπόδια. και θα βοηθηθούν οι διοργανωτές αν το τρίτο παράρτημα που θα συμπληρώνεται με προσωπικά στοιχεία ε, μαζί με τις υπογραφές να πλουστευτεί και να εναρμονιστεί όσο γίνεται περισσότερο. Να είμαστε ρεαλιστές. Πιστεύω ότι αν εξυπηρετούμε πολίτες εδώ θα πρέπει να ακούμε και τις ανησυχίες τους. Ήδη λοιπόν ε, το Κοινοβούλιο ε, τα ε, ζήτησε να γίνουν ρυθμίσεις που δυσκόλεψαν κάποια κράτη-μέλη ήδη όταν κάναμε τις διαπραγματεύσεις. Τώρα περισσότερα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να διαευκολύνουν και να εναρμονίσουν περισσότερο τη διαδικασία. Γενικά, όταν πρόκειται για συλλογή δηλώσεων υποστήριξης, το κλειδί είναι να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ προστασίας των δεδομένων και της φιλικότητας προς το χρήστη. Υπογραμμίζω και χαιρετίζω την προσπάθεια της Κομισιόν μέχρι τώρα, όπως την απόφαση να επεκτείνουν το, την προθεσμία ε, συλλογής υπογραφών για την πρώτη πρωτοβουλία. Ε, γιατί θα ήταν η πρώτη ευκαιρία που θα δινόταν. Μπορεί να ε, χρειαστεί να βελτιώσουμε, να, να φροντίσουμε ώστε οι διοργανωτές να είναι από την πρώτη μέρα έτοιμοι και να μην χάνεται χρόνος. Πολλά μπορεί να γίνουν πριν κάνουμε την αναθεώρηση του κανονισμού το 2015, διατήρηση και ενίσχυση διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή να λάβουμε υπόψη τις εμπειρίες που υπάρχουν και να ανοίξουμε μια συζήτηση για τις συγκεντρωποιημένες κεντρικές διαδικασίες. Επίσης, πρέπει να μειώσουμε στο βαθμό του δυνατού το κόστος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας. Πόσα ε, γραφεία του Κοινοβουλίου έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Πόσες δραστηριότητες διοργανώθηκαν από τα γραφεία μας. Ήταν, είμαστε ανοιχτοί στο κοινό για να συζητηθούν τα σημαντικά θέματα που τίθενται. Και για την επικοινωνία δύο θέματα είναι σημαντικά, πιστεύουμε. Το πρώτο αφορά την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών και την πρακτική χρήση της, η χρησιμότητα των ε, γραφείων ε, συνίσταται στην κοινή δουλειά γιατί πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν το νέο εργαλείο. Τώρα έχουμε ε, κάνει και κάποια καρτούν που εξηγούμε τα της πρωτοβουλίας και πώς χρησιμοποιείται το νέο εργαλείο. θα πρέπει να δούμε ε, και το θέμα των πρωτοβουλειών που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κομισιόν. Αυτό δημιουργεί απογοήτευση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που πρέπει να υπάρχουν σε ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο και θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και να δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και βοήθεια ε, ε, νομική βάση κλπ. Επίσης να υπογραμμίσω την σημασία της δημόσιας ακρόασης που την αναφέρατε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικό, ένα δυναμικό μήνυμα θα περάσει αν μπορέσουμε να το κάνουμε το Ιανουάριο εδώ στο Κοινοβούλιο όπως είπατε κι εσείς για τις επιτυχείς πρωτοβουλίες. Αυτές οι ακροάσεις μαζί με το νομοθετικό follow-up συνέχιση ε, αναδεικνύουν τις πρωτοβουλίες των πολιτών στην Ευρώπη και δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να κάνουν ανοιχτές συζητήσεις. Οι προσδοκίες των πολιτών είναι υψηλές, μεγάλες και θα πρέπει κάπως να τις ε, ε, αντιμετωπίσουμε. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, για να... οι προσπάθειές μας πρέπει να στοχεύουν οι πρωτοβουλίες αυτές να ε, αποτελέσουν ε, μια σημαντική διάσταση της δημοκρατίας. Εγώ ελπίζω ότι η δουλειά μας δεν ε, έγινε επιματέο, κρίνοντας εκ του ναι. αποτελέσματος και ευχαριστώ και πάλι εσάς κύριε Επίτροπε και την ομάδα σας. και βλέπω και άλλους συναδέλφους σας από την Επιτροπή να παρευρίσκονται. Ο κύριος Μέσος μην το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Επίτροπε, είπατε ότι εγκρίθηκαν 21 πρωτοβουλίε. Απορρίφθηκαν κάποιε. Μπορείτε να μας το πείτε. Και για ποιου λόγου, Θυμάμαι ότι εδώ είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για τους πολιτικούς λόγους ε, απόρριψης πρωτοβουλίας πολιτών θέλετε να μας τα εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Μετά, αυτοί που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, είπατε ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να ξεκινήσει ένας διάλογος με τους πολίτες της Ευρώπης. Εμείς ε, είπαμε ότι δεν θα έπρεπε πολιτικά κόμματα να εργοποιούνται στις δραστηριότητες αυτές, αλλά όχι πολιτικές οργανώσεις που δεν είναι κόμματα. Τι οργανώσεις λοιπόν ε, βρίσκονται πίσω από τις πρωτοβουλίες αυτές, ακόμα και από τις μη παραδεκτές. Υπάρχουν νέοι δρόντες ε, στο παιχνίδι ή είναι η συνήθιση ύποπτη, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αυτοί που αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, αυτοί που πάντα είχαν εμπλακεί στον ευρωπαϊκό διάλογο και βρίσκουν ένα νέο τρόπο να περάσουν τα πολιτικά τους μηνύματα υπάρχει πραγματική εμπλοκή ατόμων που στο παρελθόν δεν θα είχαν μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέπφλιν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Μου πάρα πολύ η περιγραφή της, αυτής, ε, του ξεκινήματος της δύσκολης αυτής διαδικασίας. Και από ό,τι κατάλαβα, η Επιτροπή, από αυτά που είπατε, η Επιτροπή θεώρησε ότι μπορεί να κατευθύνει το εργαλείο αυτό με έναν ευλογό τρόπο. Και έχω πολλές ερωτήσεις. Κάποιες συνδέονται με ερωτήσεις που ήδη λάβατε. Η σερβερ που είπατε ότι διαθέσατε, ήταν σερβερ προσωρινή ή μόνιμη. Γιατί στην πρώτη περίπτωση μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε να υπάρξει κάποιο κονδύλι για την μονιμοποίηση αυτών των σερβερ. Δεύτερον, τα προηγούμενα. Μιλήσατε, αναφέρατε 21 πρωτοβουλίες. Τα κριτήρια αξιολόγησης τους από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν ήδη. Και πραγματικά θα με άφηνα αποσβολωμένο αν καταφέρατε να μου δώσετε μια εικόνα από ποιους γίνεται η αξιολόγηση, είναι εξωτερική από την Επιτροπή, πώς δημιουργήθηκαν τα κριτήρια που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση. Κάποιος τα, τα έβγαλε από το μυαλό του, μια Επιτροπή τα έβγαλε από το μυαλό της. Πώς ε, έγιναν, διότι πρόκειται για το ξεκίνημα ενός νέου θεσμικού εργαλείου. Οι αποφάσεις που λαμβάνετε τώρα θα λειτουργήσουν ως προηγούμενο και μπούσολες για το μέλλον, περιορίζοντας την εμβέλεια και το πεδίο εφαρμογή της ε, πρωτοβουλίας. Επόμενο ερώτημα. Ξέρετε ποια είναι τα κράτη-μέλη, αλλά η ερώτηση που θέτω είναι οι υπογράφοντες και υπογραφές είναι διάσπαρτες μεταξύ των κρατών Υπάρχουν ε, κάποιες χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανταπροσωπευτικότητα, άλλες χώρες όπου οι πολίτες δεν πολύ ενδιαφέρονται. Πώς γίνεται η κατανομή βάσει του μεγέθους του κράτους. Οι πληροφορίε που θα μα δώσετε θα ήταν πάντα ευπρόσδεκτες. Επίσης αναφερθήκατε σε μια, στην του Ιανουαρίου. Βεβαίω πρέπει να το δούμε σοβαρό αυτό. Μιλήσατε για το δικαίωμα στο νερό. Πόσες ακροάσεις σκέφτεστε να οργανώσετε στο εγγύς μέλλον ή τέλο πάντων έχουν ξεκινήσει. Διότι ξέρετε ότι έχουμε εκλογές σε λίγο. Οι εκλογές σίγουρα θα μειώσουν την προσοχή σε μια ακρόαση που είναι σημαντικό, που είναι σημαντικές για την επίγνωση του πολίτη. Η ερώτησή μου είναι, έχετε κι άλλες ή είναι μόνο αυτοί για το νερό. Γιατί θα κάτσουν πάνω στις, ε, στην προεκλογική εξτρατεία που δεν είναι κάτι καλό. Να κλείσω ακολουθώντας και αυτά που είπε η κυρία Γκουρμάη για τα γραφεία του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε πληροφορία έχουμε για το θέμα αυτό θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Επίσης θέλω να ξέρω σε τι βαθμό, αν υπάρχει, ε, λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο περιφερειακών γραφείων. Ε, εντάξει, εσείς είστε από μικρή χώρα, αλλά και πάλι και στην, μπορεί, μπορεί να θέλετε να βάλετε και ένα γραφείο στο Κόσιτσε, για παράδειγμα, πέραν της Μπρατισλάβα, αλλά σε άλλες χώρες με τα ελιώτικα. Έχετε στο Εδιμβούργο, τι γίνεται, τι γίνεται στην Ισπανία. Θα ήθελα να έχω μια καλή εικόνα της περιφερειακής διάστασης των ε, γραφείων, γιατί βέβαια όσο πιο κοντά στον κόσμο είναι η πρωτοβουλία τόσο πιο απτή για τον πολίτη είναι. Ο κύριος Νταφ. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα. Τρεις έχουν ολοκληρωθεί. Και επίκειται η πιστοποίηση από τις εθνικές αρχές. Μία είναι για το δικαίωμα του δημοσίου τομέα να ελέγχει τις υπηρεσίες υδάτων και πολύ θα ήθελα παρακαλώ να μας πείτε περισσότερα πράγματα για την ουσία αυτών των τριών. Ε, η πρώτη υποστηρίχθηκε από τη συνδικάτα του δημοσίου τομέα που ήταν κατά της ε, ιδιωτικοποίησης ε, των εταιριών ύδατος. Η δεύτερη για τις αμβλώσεις, που φαντάζομαι ότι είναι κατά των αμβλώσεων και προωθούνται από την Εκκλησία, για να απαντήσω κιόλα στον κύριο Μέσερ Σμιτ. Και η τρίτη είναι για τα πειράματα στα ζώα, για ιατρικούς σκοπούς. Πίσω από αυτήν είναι οι ομάδες ε, που είναι κατά των πειραμάτων στα ζώα και υπέρ της καλής κατάστασης των ζώων. Αυτά όλα είναι οριακά σε σχέση με τις ενωσιακές ε, αρμοδιότητες. Μπορεί να ερμηνεύσουμε εκτατικά ε, το θέμα και να πούμε ναι, είναι θέματα αυτά για τα οποία μπορεί να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, για την καλή κατάσταση των ζώων, ήδη έχουμε οδηγία για την καλή τους διαβίωση κλπ που καλύπτει και την χρήση ζώων στην ιατρική έρευνα. Ε, τώρα, εγώ πέρα από την επιβεβαίωση που θέλω από εσά, σχετικά με αυτά που είπα, ερωτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα σχέδιο της αιτιολογημένης γνώμης της ε, πριν από τη δημόσια ακρόαση για όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει την ε, δημόσια συζήτηση και θα γίνει πιο στοχευμένη η συζήτηση στις ακροάσεις που θα κάνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι έτοιμη τότε που θα γίνουν οι ακροάσεις να παρουσιάσει τις πρώτες της σκέψεις σχετικά με την επιλεξιμότητα όλων αυτών των πρωτοβουλειών με βάση τις αρμοδιότητες που προβλέπει η συνθήκη. Ευχαριστώ κύριε Σέφνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάντοτε χαρά να σας βλέπουμε εδώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Το Σεπτέμβριο όταν ε, Μιλήσαμε για την μικρή μεταρρύθμιση στα πλαίσια της μιας κατεξουσιοδότηση πράξης. Προτείναμε το, να προχωρήσουμε χωρίς ε, πρόβλημα, αλλά να κάνουμε μια συζήτηση και με εσά και με το Συμβούλιο. Και λυπάμαι που δεν εκπροσωπείται η Προεδρία του Συμβουλίου. Γιατί καλό είναι να κάνουμε έναν απολογισμό τώρα και να δούμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, τι χρήζει βελτίωση, Και πρέπει να πω ότι το μεγάλο αυτό καινούριο μέσο, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, επιτρέπει στους πολίτες για πρώτη φορά απευθείας να ε, θέτουν θέματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λένε ότι θέλουμε να γίνει κάτι σε αυτό το τομέα, να βελτιωθεί κάτι κλπ. κλπ. Αυτό είναι μεγάλο βήμα, μεγάλη βελτίωση. Και ήταν ένα εντελώς καινούριο βήμα. Δεν υπήρχε προηγούμενο εδώ και διαπιστώνουμε ότι εν μέρη πετύχαμε, εν μέρη οι προσδοκίες δεν δικαιώθηκαν. Εν μέρη υπήρχαν και οργανωτικά και τεχνικά προβλήματα που δεν τα είχαμε προβλέψει και εσείς που είστε υπεύθυνοι για αυτό το εγχείρημα που συμμετείχατε και στη διαμόρφωση του κανονισμού και εμείς ε, μαζί θα έχουμε την ευθύνη να δούμε τι ε, πήγε καλά και τι όχι και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Νομίζω και αναφέρομαι εδώ σε αυτό που είπε ο Άντριου Νταφ, ότι ε, το ένα εκατομμύριο υπογραφές και τα όρια που δημιουργήσαμε με τη συλλογή υπογραφών στα κράτη-μέλη, ε, αυτός ο αριθμός δεν πιάνεται εύκολα και οι πρωτοβουλίες που δεν έχουν μια καλή οργάνωση δυσκολεύονται πολύ. Ε, μέχρι τώρα είχαμε λίγες πρωτοβουλίες, τρεις, που ανταποκρίθηκαν στον πύχη που είχαμε θέσει. Γιατί από πίσω κρύβονται ισχυρές, ισχυροί διοργανωτές. Είχαμε και άλλες πρωτοβουλίες, άλλες πρωτοβουλίες χωρίς μεγάλη και γερή ε, οργανωτική βάση που άρχισαν από πρωτοβουλίες πολιτών, κάποιες οργανώσεις και άμα δούμε τις ε, συλλογές των υπογραφών βλέπουμε κάποιες χιλιάδες, καμιά φορά δεκάδες χιλιάδες, αλλά πολύ λιγότερες. Και όλοι οι υπεύθυνοι νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν ότι ο μεγάλος στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα μέσον ώστε και εκείνοι που δεν έχουν γερό οργανωτικό μηχανισμό και εκείνοι να μπορούν να ε, θέτουν με αποτελεσματικό τρόπο ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό εν μέρη το πετύχαμε. Και αν πρέπει να ξανασκεφτούμε κάτι πρέπει να σκεφτούμε να διευκολύνουμε τα πράγματα, όχι να τα ε, περιπλέξουμε περισσότερο. Τώρα, οι πολλές μεγάλες τεχνικές δυσκολίες. Εδώ θα πρέπει να ε, δούμε εμείς τι κάνουμε. Μέχρι τώρα το προωθήσαμε, το προβάλαμε στους πολίτες, αλλά δεν φροντίσαμε να λειτουργεί όπως πρέπει. Επί μισό χρόνο αφήσαμε να ταλαιπωρούνται οι πολίτες από τεχνικές δυσκολίες. Κάποιοι κουράστηκαν και σταμάτησαν, ε, άλλοι έπρεπε να ε, βοηθηθούν να ε, προσφύγουν σε άλλες εταιρείες. Αυτό δεν ήταν καλή αρχή πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα. Πρώτον, και το συνδέω αυτό με μία ερώτηση προς εσάς. Ε, αποφασίσατε και σας ευχαριστούμε την προθεσμία να την παρατείνετε ή να την ξανααρχίσετε, να αρχίσει πάλι να τρέχει. Και έχουμε και αυτή τη λύση ad hoc για τον σερβερ στο Λουξεμβούργο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η λύση θα είναι λειτουργική, αλλά δεν είναι μία λύση που αναφέραμε ως ε, στάνταρ. Είναι μια λύση προσωρινή. Όμως ε, θα πρέπει να είναι σαφές πώς θα τρέξουν οι άλλες πρωτοβουλίες κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις ή όχι. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε ένα μέτρο να το προβλέπουμε για ορισμένες πρωτοβουλίες και για ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά είναι ισχύει για όλες. Δεύτερον, Έχω την εντύπωση ότι πολλές τεχνικές δυσκολίες οφείλονται στο ότι δεν είχε γίνει αρκετά μακροπρόθεσμος και σωστός σχεδιασμός. Ε, οι διαδικασίες των δοκιμών που συνήθως τρέχουν ε, σε τέτοια συστήματα πριν αυτά τεθούν ε, σε κοινή λειτουργία, όλα αυτά δεν είχαν γίνει. Κάποια λάθη μπορούσαν να αποφευχθούν. Υπήρχαν όμως και πολλά προβλήματα τα οποία απορρέουν από τον ίδιο τον κανονισμό. Εμείς θέλαμε πάντοτε και εγώ συμφωνώ σε αυτό μαζί σας κύριε Σεύκοβιτς. Πάντοτε λοιπόν θέλαμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο και για τις υπογραφές των πολιτών. Δηλαδή αυτή είναι ευρωπαϊκή και όχι εθνική πρωτοβουλία των πολιτών και η επιθυμία μας ήταν να μπορούμε να λέμε όνομα διεύθυνση, Ξέρουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη χρειάζεται και ε, τόπος και ημερομηνία γέννησης. Αρκούν αυτά για να βάλει κανείς εγγράφο στην υπογραφή του ε, ή με το διαδίκτυο και να υπάρχει επαλήθευση. Υπάρχει το πρόσωπο, ε, επαληθεύουμε έτσι, ότι υπάρχει το πρόσωπο και υπέγραψε μία φορά. Τώρα, το μεγαλύτερο λάθος, θα με συγχωρήσετε που το λέω, το μεγαλύτερο λάθος της Κομισιόν ήταν η επιστολή προς τις διοικήσεις των κρατών μελών που τους ρωτήσατε τι έγγραφα θέλετε για την επαλήθευση. Αυτό ε, δημιούργησε αντανακλαστικά. Με ελάχιστες εξαιρέσεις τα κράτη-μέλη ανέφεραν έγγραφα. Η Γερμανία είπε θέλουμε ταυτότητα και διαβατήριο. Ενώ αυτό δεν αληθεύει γιατί στη Γερμανία έχουμε πολύ πιο νομικά δεσμευτικά ε, μέσα για τους πολίτες ε, μέχρι πρωτοβουλίες ε, και δημοψηφίσματα μπορεί να αλλάξουν και την νομοθεσία. Και παντού βάζουν μόνο υπογραφή, όνομα, διεύθυνση. αυτό το επιβεβαίωσε και, το, και για το Κοινοβούλιο και ο, ο συνήγορος του πολίτη. Αυτό δεν έπρεπε. Η Κομισιόν ρώτησε. από τη Γαλλία είπαν 18 έγγραφα για να είναι σίγουροι. Άλλοι είπαν ένα, άλλοι είπαν τέσσερα. Κομικό. Τώρα καταφέραμε κάποια κράτη-μέλη να μην ζητάνε τα έγγραφα, αλλά όμως όχι. Και έχουμε ένα μακρό κατάλογο και κάπως με την κατεξουσιοδότηση πράξη το διορθώσαμε λίγο αυτό, βραχύναμε λίγο τον κατάλογο, αλλά πάντως υπάρχει κατάλογος. Και ε, μια σειρά κρατών μελών βάζει δικά τους κριτήρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν, μπορούν, δεν θα υπογράφουν πολίτες, αλλά το πρώτο που πρέπει να πούνε είναι είμαι Γάλλος, είμαι Άγγλος, είμαι Πορτογάλος και μετά αρχίζει να τρέχει στο background μια άλλη σελίδα και έρχεται με πρόσθετες ερωτήσεις. Αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαράδεκτο. Η ιστοσελίδα είναι πολύ περίπλοκη και μπερδεύει και τους πολίτες. Ε, βάλαμε μια προθεσμία μέχρι το 2015 για να τα μεταρρυθμίσουμε αυτά. Και αν θέλουμε να το κάνουμε το 2015 πρέπει να αρχίσουμε τώρα συνομιλίες με τα κράτη-μέλη και να τους πούμε μπορείτε να φροντίσετε σε κάθε χώρα να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα και να μπορούν να υπογράφουν υπό τις ίδιες συνθήκες ανεξάρτητα από που μένουν. Τώρα υπάρχουν 11 εκατομμύρια στην Ευρώπη που δεν μπορούν να υπογράψουν γιατί μένουν σε άλλη χώρα από τη χώρα που έχουν την ηθαγένεια κλπ. Αυτό σε εθνικές εκλογές μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Και αυτό λύνεται. Αλλά δεν μπορεί να είναι πρόβλημα σε αυ... εν, προκειμένου. Και θέλω να μου πει η Κομισιόν και το Συμβούλιο πάνω από όλους, γιατί εκεί ε, βρίσκεται το πρόβλημα, αυτή είναι η αρμόδια και κρίμα που δεν είναι εδώ, να μας πει το Συμβούλιο τι πρέπει να γίνει τόσο ώστε το μέσο συμμετοχής των πολιτών να απαλλαγεί από τα εμπόδια που έχει και να γίνει ένα ευρωπαϊκό μέσο φιλικό για τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως το είχαμε ευθύ εξ αρχής φανταστεί. Τέλος μια ερώτηση ακόμη. Εγώ από την αρχή είχα εκφράσει την ανησυχία ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε κάποιους συνεργάτες, πολύ αφοσιωμένους, ενθουσιώδεις, αλλά δεν είναι αρκετός ο αριθμός τους. Όλες οι, όλα τα, οι καταγγελίες που φτάνουν σε μένα μέσα από τις πρωτοβουλίες και πολλές φορές ε, εκφράζουν ε, καταγγελίες και παράπονα, όλα αυτά δείχνουν ότι το προσωπικό που διατίθεται αλλά και οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στο νέο αυτό μέσον. Σας ερωτώ λοιπόν, τι σχέδια έχετε για το μέλλον, θα αυξήσετε τα κονδύλια και το προσωπικό. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα ε, σε αυτά τα πλαίσια. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ο Μάριο Τενρέρο, εξαιρετικός συνεργάτης, ο οποίος πολλές φορές ήρθε και μας ενημέρωσε. Του χρωστάμε πολλά ε, γιατί εκείνος δούλεψε με μεγάλη αφοσίωση και δυναμισμό και φρόντισε να λυθούν πολλά προβλήματα. Ήταν πάντοτε στη διάθεσή μας και πάντοτε πρόθυμος να βρει λύσεις ε, και με τα κράτη-μέλη. Και τον ευχαριστώ θερμά για τη δουλειά που έκανε. Ρωτώ όμως παράλληλα, γιατί στην Κομισιόν ελήφθη η απόφαση η ευθύνη για τις πρωτοβουλίες να μην βρίσκονται πια στα χέρια του Μάρκο Τενρέρο, αλλά να τις αναλάβει άλλος. Αυτό είναι κατανόητο για μας που παρακολουθήσαμε το θέμα, γιατί ο Μάριο ήταν εγγύηση επιτυχίας. Ε, έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν θα τις πω όλες τώρα. Μπορώ και γραπτός να στείλω, να μην μακρηγορήσω, αλλά ε, στις ερωτήσεις που σας έκανα παρακαλώ να μου απαντήσετε, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε το μέσο που προσφέραμε, ώστε οι πολίτες να συμμετέχουν και να εκφράζουν τη γνώμη τους για τα ευρωπαϊκά θέματα και να μην εμποδίζονται από τεχνοκρατικά, γραφειοκρατικά και νομικιστικά προβλήματα. Ευχαριστώ, κυρία Λένκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεκτική προσέγγιση που ακολουθείτε πάνω σε αυτό το πολύτιμο δημοκρατικό εργαλείο, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ελπίζω το δικαίωμα των σεξουαλικών μειονοτήτων, εθνικών μειονοτήτων, όπως πρόσφατα στην κρατία ελπίζω να μην το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Πολιτών, αλλά θα ήθελα τώρα να συζητήσω λίγο περαιτέρω τα περί πρωτοβουλίας πολιτών και να θέσω ένα ερώτημα σε δύο μέρη. Πρώτα απ' όλα, τη φιλικότητα προς το χρήστη, πώς τη βελτιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα τεχνικά ζητήματα φιλικών προς το χρήστη δικτύων. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο προέκυψε αφού του τέθηκε σε ισχύ η πρωτοβουλία των πολιτών. Και δεύτερο ερώτημα, όπως είπε ο επικεφαλής μονάδας για τα γενικά θεσμικά θέματα της Επιτροπής στη συνεδρία της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την πρωτοβουλία των πολιτών το Σεπτέμβριο. Παρά τις προσπάθειες Κομισιόν να εξηγήσει τους κανόνες πρωτοβουλίας των πολιτών, πολλά αιτήματα καταχώρησης έπρεπε να απορριφθούν λόγω του ότι ήταν προδήλωση εκτός ε, των εξουσιών ε, εργοδοτήτων της Κομισιόν τα θέματα των πρωτοβουλίων ε, των πολιτών. Αυτό είναι η παραποπή και σας ρωτώ με δυνάμει των συνθηκών πόσες πρωτοβουλίες πολιτών αναγκαστικά δεν απορρίψετε. Τώρα ο κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα Υπάρχει ένα μπέδεμα με τα ονοματεπώνυμα στα κροατικά μεταξύ του συναδέλφου μίλησε προηγουμένως και εμένα, αλλά τέλος πάντων. Ξέρω ότι ο κύριος Εύκοβιτς καταλαβαίνει τα κροατικά μια χαρά. Τα έχουμε ήδη πει και στο κροατικό κοινοβούλιο. Δύο ερωτήσεις θέλω να θέσω. Πρώτον, εξαιρετική, εξαιρετικό εργαλείο συμμετοχής η πρωτοβουλία πολιτών για την νομοθετική διαδικασία στις Ευρω... στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε μια σειρά θεμάτων. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε νομοθετικά κείμενα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι έδειξαν ήδη το ενδιαφέρον της Επιτροπής μας κυρίως για τα μεθοδολογικά ζητήματα. Το άρθρο 10.1 γ ιδίως, τον τρόπο με τον οποίο Δηλαδή η Επιτροπή αποφασίζει διαδικαστικά αν θα δεχθεί ή όχι μία πρωτοβουλία πολιτών. Αυτό είναι καθοριστικό για το μέλλον ε, του μηχανισμού. Πέραν του ότι αν ένα το ένα εκατομμύριο υπογραφές είναι πολλές ή λίγοι. Η Κροατία είναι μια μικρή χώρα και παρόλα αυτά έχουμε ξεκινήσει δύο πρωτοβουλίες έχοντας μαζέψει 600.000 για τη μία και 700.000 υπογραφέ για την άλλη. Μια χώρα μικρή επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω σε σχέση με την Ευρώπη ε, των 500 εκατομμυρίων. Το 1 εκατομμύριο δεν είναι εύκολο να πετύχουμε, δεν είναι εύκολο νούμερο. Κατόπιν θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα γραφεία που βρίσκονται σε κρατικό επίπεδο, σε κρατημέλη. Τα γραφεία δηλαδή που υπάρχουν ε, στα κρατη και συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών. Στην Κροατία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα γραφείο σωματείων που ασχολείται δηλαδή με την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Θα μπορούσε να βοηθήσει την Κομισιόν Μπορεί λοιπόν η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες αυτές και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με την συμμετοχή στις ε, κοινοβουλευτικές ευρωεκλογέ που έχουμε. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα θετική πρωτοβουλία και πρέπει να βελτιώσουμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πρόκειται για νέα πρωτοβουλία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε την πρωτοβουλία αυτή και θα δούμε αν καταφέρουμε να προωθήσουμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Έφνερ που ζήτησε το λόγο ξανά, θέλω και εγώ να ζητήσω από τον εδώ κάποιε διευκρινήσει και να του κάνω και κάποιε προτάσει. Φερρυπίν. Όλοι ρωτήσανε ο σερβερ είναι μόνιμος ή όχι. Καθοριστική σημασία. Πάντως, εφόσον μιλούμε για αλλαγή, πιθανή αλλαγή του κανονισμού, η σύμπτωση μεταξύ της στιγμής καταχώρησης και της στιγμής της πιστοποίησης του, email πρέπει να αλλάξει. Ε, λέει αυτή τη στιγμή ο κανονισμός οι υπογραφές αρχίζουν να συλλέγονται μετά την καταχώρηση. Ενώ ε, μετά λέει ότι δεν μπορεί να λαμβάνονται τα email πριν την πιστοποίηση. Θα έπρεπε λοιπόν να Ε, διαμορφωθεί, να αναδιαμορφωθεί το κείμενο, το κείμενο εκτός αν ας πούμε η οργάνωση που ξεκινάει τη διαδικασία συλλογής υπογραφών λέει θα το κάνω μόνο επί χάρτου. Επίσης ο κανονισμός προβλέπει επαφή των οργανωτών της πρωτοβουλίας με την Επιτροπή. Η εμπειρία θα δείξει κατόπιν τι νομοθετικές ρυθμίσεις απαιτούνται στο μέλλον. Η ερώτηση ωστόσο είναι από την Οργανωτική Επιτροπή ποιος θα έχει την επαφή. Τα άτομα που αναφέρονται την πρόταση που δεν μπορεί να είναι πάνω από 7, αλλά η επιτροπή μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Άλλοι εμπειρογνώμονε θα συνοδεύουν ή όχι, πώ σε ποιο πλαίσιο. Επίτροπο, υπάλληλο, ομάδα επιτρόπων, ολόκληρη την επιτροπή. Τρίτον, με τι αποτελέσματα. Ο κανονισμός λέει ότι οι διοργανωτέ μπορούν, μπορούν όχι οφείλουν, να διατυπώσουν και νομικό κείμενο. Κάποιοι το έκαναν, άλλοι δεν νομίζω το έκαναν. Σε τι βαθμό η συζήτηση μπαίνει στη διατύπωση. Αν δεν υπάρχει διατύπωση, είναι άλλη περίπτωση. Θα επανέλθω και σε αυτά που είπε ο κύριος Νταφ. Η καταχώρηση προϋποθέτει ότι υπάρχει αρμοδιότητα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι άπαξ και καταχωρηθεί ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται μπορεί η Επιτροπή να πει ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας. Από τη στιγμή που γίνεται καταχώρηση ε, υπάρχει αρμοδιότητα. Μπορεί να μην υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Άλλη ερώτηση. Ποιος προτείνεται για συνομιλητής, ένα άτομο, η Επιτροπή ή κάποιος προτείνει Επιτροπή. Επίσης, ο κανονισμός λέει τους επόμενους τρεις μήνες, αλλά οι τρεις μήνες μπορεί να πέσουν στο, στην περίοδο της προεκλογικής εξαρτίας. Καλοκαίρι. Μήπως πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν μια παράταση του τρίμηνου είναι άκαμπτος δεσμευτικός ο κανόνας. Είναι δηλαδή ενδεικτική ή υποχρεωτική η προθεσμία. Αυτό είναι σημαντικό και εν ώψη της πιθανής αναθεώρησης του κανονισμού. Θέλει κάτι ακόμα ο Χέφνερ, αλλά σύντομα παρακαλώ. Σύντομα, σύντομα για το ίδιο θέμα. Πολύ σύντομα θα γίνει η πρώτη ακρόαση. Και είπατε ότι προτείνεται να γίνει τον Ιανουάριο. Από ό,τι γνωρίζω, λίγες προετοιμασίες έχουν γίνει. Η ακρόαση Είναι ένας τρόπος να ε, προωθήσουν το δίκαιο αίτημά τους οι διοργανωτές με τις υπογραφές. Και ε, εκείνοι που εργάζονται πάνω σε αυτό το θέμα και εγώ που μιλάω με όλους τους άλλους ε, εμείς λοιπόν μέχρι τώρα δεν είχαμε συμμετάσχει στη διοργάνωση αυτών των ε, ε ακροάσεων και ανησυχώ και περισσότερο αν προχωράμε σωστά. Ε, για παράδειγμα είχαμε πει να υπάρχει μια επιτροπή πρωτοβουλίας με 7 άτομα από 7 χώρες. Και είχα καταλάβει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι τουλάχιστον αυτή η Επιτροπή Πρωτοβουλίας θα έπρεπε να προσκληθεί και ίσως και δυο-τρεις εμπειρογνώμονες που θα ορίζονταν. Ε, βλέπω τώρα ότι δεν καλύπτεται το κόστος ταξιδίου των μελών της Επιτροπής ε, Πρωτοβουλίας. Οπότε κάτι που πήγε καλά, άρχισε καλά πάει τώρα να κολλήσει μέσα από μια μικρόψυχη απόφαση. αφού λοιπόν είχαμε ε, θεσπίσει νομικά επταμελή επιτροπή πρωτοβουλίας, όχι πρόεδρους και αντιπροέδρους, όλοι ισότιμοι είναι. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον οι 7 αυτοί να προσκληθούν και να συμμετέχουν στην ακρόαση και να μιλήσουν και εκείνοι. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συζητήσεις αυτές πώς θα οργανώσει τη δική της τη συμμετοχή. όπω ας πούμε το δικαίωμα στο νερό και θα εξηγήσει, πώς θα εξηγήσει ότι ε, υπάρχουν ε, τρεις διαφορετικοί τομείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Στο σχέδιο για την ε, επανεξέταση το 2005 θα πρέπει να έχουν στηριχθεί σε όλες αυτές τις εμπειρίες. Ευχαριστώ. Κάμποσες παρεμβάσεις. Το λόγο έχει τώρα ο Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για τις ε, ερωτήσεις τους και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για αυτό το εξαιρετικά πολύπλοκο και σημαντικό θέμα. Η υποστήριξη και η ε, στο ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ε, για πρώτη φορά ήταν πολύ χρήσιμε. Δεν θα απαντήσω σε κάθε μία ερώτηση χωριστά, θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω κάποιες. Ξεκινώ με την εισηγήτρια κυρία Γκουρμάη. Η ερώτησή τη για την αναθεώρηση αντικατοπτρίζει κάποια από τα θέματα που έφυγε και ο κύριο Χέφνερ και η κυρία Πέτροβιτς Ιακοβίνα. Είναι σαφές ότι αφού περάσει, ολοκληρώσουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο το Μάρτιο φέτος, θα έχετε αρκετέ πληροφορίες για να, για να προετοιμάσουμε την επόμενη αναθεώρηση. Βεβαίω αυτό θα είναι θέμα του επόμενου Κοινοβουλίου και της επόμενης Επιτροπής μπορώ να σας πω την άποψή μου για το τι νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε για να καταστήσουμε τη διαδικασία ευκολότερη, φιλικότερη στον πολίτη και να ε, αυξήσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών για την πρωτοβουλία. Να πω καταρχάς την κυρία Γκουρμάη και τον κύριο Σαφλίν ότι πρέπει να απλοποιήσουμε περαιτέρω τις απαιτήσει δεδομένων σε ό,τι αφορά την υπογραφή ή την υποστήριξη πρωτοβουλία. Επίσης να σας πω ότι χαίρο που βλέπω ότι ήδη σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν θετικά μηνύματα από τα κράτη-μέλη που προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό των στοιχείων που απαιτούν από τους πολίτες και να αντιμετωπίσουν κάποια από τα θέματα που ανέφερε ο κύριος Χέφνερ. ότι υπάρχουν περίπου 11 εκατομμύρια πολιτών που δεν μπορούν να συμμετάσχουν λόγω προβλήματος ε, επίσημης κατοικίας τους. Έχουμε ένα πρόβλημα, έχουμε ένα θέμα, μια περίπτωση θετική στην Ολλανδία που έλυσε το ζήτημα είναι αλλαγή στη φόρμα που χρησιμοποιούν οι πολίτες, οι Ολλανδοί πολίτες και επιτρέποντας έτσι σε Ολλανδούς πολίτες που δεν μένουν στην Ολλανδία που δεν έχουν την κατοικία τους δηλαδή στην Ολλανδία εκείνη τη στιγμή να δείξουν την υποστήριξή τους για μια πρωτοβουλία. Είναι εφικτό λοιπόν και νομίζω ότι πρέπει να διδαχθούμε από τα θετικά παραδείγματα και να προσπαθήσουμε να τα διευρύνουμε σε όλα τα κρατημέλη. Νομίζω ότι στο ξεκίνημα υπήρχε κάποια ανησυχία για το διοικητικό άχθος, το πόσο μεγάλη θα ήταν η διαδικασία αυτή, το πώς θα αντέχαν πως ανταποκρίνονται τα κρατημέλη στις απαιτήσει της επαλήθευση, αλλά όταν, το... ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή η ταυτοποίηση, είδαμε ότι δεν υπήρχαν μείζωνα προβλήματα στα κράτη-μέλη, ενώ κατάλαβαν ότι δεν και κάτι το ασύλληπτα περίπλοκο. Εμείς κάναμε τυχαίους ελέγχους, και από αυτό κάναμε αναγωγές αποτελεσμάτων. Δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι είναι ε, 1.321.241 πολίτες, απλά ότι είναι μια πραγματική ουσιαστική πρωτοβουλία, ότι οι άνθρωποι είναι όντως άνθρωποι και τα νούμερα είναι αντίστοιχα. Αυτό θα επιτρέψει περαιτέρω απλοποίηση των παρατημάτων επίσης θα λειτουργήσει, θα πάψει να είναι αποτρεπτικό για τους πολίτες, δηλαδή οι οποίοι βλέπουν ε, το έντυπο και λένε πρέπει να τα συμπληρώσω όλα αυτά και να τα δώσω σε κάποιο μηχάνημα. Η απλοποίηση των παρατημάτων θα επιτρέψει να πετύχουμε πολλά. Δεύτερο θέμα. Και χρησιμοποιώ τις ιδέε που συζητήσαμε στις βασικέ συζητήσει, δυστυχώ όμω τότε λίγοι, πολύ λίγοι ήταν αυτοί που μπορούσαν να το σκεφτούν αυτό. Στο μέλλον, το ευκολότερο για την ε, πρωτοβουλία πολιτών θα ήταν να υπάρχει μία ενιαία θύρα πρωτοβουλίας πολιτών όπου θα υπάρχουν όλες οι πρωτοβουλίες και όλες οι πληροφορίες Ποιες πρωτοβουλίες απορρίφθηκαν, τι επιπλέον προτάσεις χρειάζονται. Βέβαια, πρέπει να έχεις ε, από πίσω έναν ισχυρό σερβερ και μια ομάδα που φροντίζει τον σερβερ για να δουλέψει σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας, όλους τους κανόνες ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα που έμαθα στις επαφές μου με τις αρχές του Λουξεμβούργου, διότι μόνο όταν μπει σε μια τέτοια λεπτομεριακή διαδικασία θα καταλάβεις τι παίζει και τι μπορεί να συμβεί όταν είσαι υπόλογος, υπεύθυνος πιο σωστά, για ένα εκατομμύρια προσωπικών δεδομένων. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ευκολότερο να το χειρίζονται ευρωπαϊκά όργανα, αλλά με το σωστό προπολογισμό, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ευτυχώ είμαι υπεύθυνο και για την πληροφορική στην Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση Digit που ήταν υπεύθυνη και οι οποίοι ήταν πολύ βοήθεια επιβοηθητικοί, επέτρεψαν να μιλήσουμε με τις αρχές του Λουξεμβούργου, που ήταν πολύ επιβοηθητικές με τη σειρά τους. Ε, κάναμε τα τεστ τζάπα γιατί αυτό στοιχίζει. Το να έχεις λοιπόν μία θηρίδα με γερό ε, σερβερ, μια σωστή ομάδα, μια καλή ομάδα και αρκετό προϋπολογισμό θα διευκολύνει την όλη διαδικασία αποφεύγοντας ε, τα τεχνικά προβληματάκια Μπορεί να γίνει έτσι. Και ξέρω ότι πολλά από όσα σας λέω προτάθηκαν και νωρίτερα, αλλά ότι ήταν δύσκολο να το δεχθούν πολλοί. Νομίζω ότι τώρα, άπαξ και ότι άμα καταλάβεις ότι δεν είναι και τόσο περίπλοκο, ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε καλύτερη επίδοση e-government. Όσοι έχουν καλή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έχουν πιο σύγχρονη διοίκηση, καλύτερη οικονομία, καλό επιχειρησιακό περιβάλλον και πιστεύω ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία θα είναι η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι νέοι ιδίω θέλουν, να είναι όλο και περισσότερο σε απευθείας επαφή με τις αρχές μέσω των email, των κοινωνικών ε, μέσων και όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε ότι οι διαβουλεύσεις στην Επιτροπή τουλάχιστον αποκτούν περισσότερο την ε, μορφή ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων. Ε, λειτουργούμε κάπως πρωτοπόρο εδώ σε ένα τομέα που μπορεί να γίνει mainstream σε λίγα χρόνια. Συμφωνώ λοιπόν με τη Ζήτα και τον Κέροντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναθεωρήσουμε και να ενημερώσουμε τις διαδικασίες για την πρωτοβουλία των πολιτών με βάση τις τελευταίες τεχνικές απαιτήσει. Τώρα, να πηδήξω στο θέμα της ακρόασης. Πολύ το έθεσαν ο πρόεδρος, ο κύριος Νταφ, η κυρία Πέτροβιτς. Something which uh, we would have to do uh, for the first time. We... Και αυτό δεν το κάναμε πρώτη φορά. Κάναμε ένα γρήγορο υπολογισμό και είδαμε ότι αν λάβουμε ηλεκτρονικά αποδεδειγμένα στοιχεία από ένα εκατομμύριο πολίτε, Περιμένουμε ακόμα τα τελικά νούμερα από δύο-τρία κράτη-μέλη. Βάσει του κανονισμού θέλουμε να, να εκδώσουμε ανακοίνωση σε τρει μήνες. 17 Μαρτίου είναι η ημερομηνία. Ζητούσε λοιπόν η ακρόαση να γίνει τον Ιανουάριο ήδη για να μπορέσουμε να περιλάβουμε την έκβα, το αποτέλεσμα της ακροασής στην ανακοίνωσή μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε, είναι, ξέρουμε ότι είναι φορτωμένη η προεκλογική εκστρατεία, και νομίζω ότι το πώς θα χειριστούμε την επικοινωνία στο τομέα αυτό είναι σημαντικό για το πώς βλέπουν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου οι πολίτες στην πρωτοβουλία πολιτών. Η οργάνωση τώρα της ακρόασης προφανώς είναι κάτι που πρέπει να, συζητηθεί ε, σημαντικά και με το Κοινοβούλιο και, και στο ιστορικό του Κοινοβουλίου πρώτα και με την Επιτροπή που θα σας βοηθήσει όσο περισσότερο γίνεται. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ε, αν δεν κάνω λάθο η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η ΕΝΒΗ είναι αυτή που θα οργανώσει την ακρόαση και ο καλύτερο νομίζω τρόπος είναι να το συζητήσουμε εσωτερικά με τους οργανωτές για το μέγεθος και τους προσκεκλημένους και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας να δεχθούμε τους οργανωτές είτε πριν είτε μετά την ακρόαση, για να μην χρειαστεί να έρθουν δύο φορές στις Βρυξέλλες. Τώρα, πόσους θα καλωσορίσουμε εκ νέου στις Βρυξέλλες, αυτό είναι κυρίως ε, απόφαση του Κοινοβουλίου και αφορούσε και το θέμα του κόστους ταξιδιού και των ε, διαδικασιών ε, οργάνωση ταξιδιού των οργανωτών και των εμπειρογνωμόνων που εσείς θέλετε να καλέσετε στις ακροάσεις. Θα ήταν σκόπιμο να το προετοιμάσουμε σωστά, θα ήταν μοντέλο και τις επόμενες ακροάσεις που πρέπει να οργανώσουμε. είχε τεθεί και το θέμα, α, το ερώτημα του κύριου Σέπλιν τώρα, πόσα τέτοια, πόσες ακροάσεις δουλεύουμε. Ε, άλλες δύο νομίζω, που περιμένουν ε, τη διαδικασία από τα κράτη-μέλη. Ε, άρα πριν της, ε, τη λήξη της θητείας σας θα έχουμε άλλες δύο μάλλον ακροάσεις. Εμείς προετοιμάζουμε τις ανακοινώσεις για τις δύο αυτές πρωτοβουλίες. Ερώτηση. Έχουμε αρκετό κόσμο ή τι σημαίνει η προετοιμασία μια τέτοια ανακοίνωση. Το δικαίωμα για το νερό είναι μια σύνθετη διαδικασία. Το ρώτησε ο κ. Νταφ. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ιδιωτικοποίηση τη εταιρεία παροχή ε, νερού, αλλά έχει και θεωρητικές διαστάσεις. Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, τι κάνει η Ένωση στον τρίτο κόσμο π.χ η δική μας λοιπόν ανάλυση δείχνει ότι, για να συντονί... ότι χρειάζεται συντονισμός ε, αποφάσεων μεταξύ επτά γενικών διευθύνσεων όπου ο συντονισμός θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία. Το πώς θα προχωρήσουμε τώρα για την έγκριση της ανακοίνωσης θα γίνει με ενδοϊπηρεσιακή διαβούλευση υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας. Και εν τέλει, λόγω και της πολιτικής σημασίας, θα εγκριθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Αυτή είναι και η συνήθιση διαδικασία τώρα για τον αριθμό των υπαλλήλων. Από ό,τι άκουσα στην πρώτη συντονιστική συνάντηση, ήταν 100 οι υπάλληλοι που ασχολήθηκαν ε, με το θέμα, που συναντήθηκαν δηλαδή, Ο κ. Μέσσερ Σμιτ με ρώτησε για τις απορρίψεις πρωτοβουλειών και η κυρία Πέτροβιτ σωστά ανέφερε το κείμενο του κανονισμού. Μπορούμε λοιπόν να απορρίψουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες μόνο που είναι προδήλως εκτός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταχρηστικές, ασήμαντες Αυτές είναι οι βασικές ε, προϋποθέσεις. Εμείς είμαστε προσεκτικοί. Πάντα η νομική υπηρεσία και η επικεφαλής γενική διεύθυνση συντονίζουν την απάντησή μας, διότι ξέρουμε ότι οποιαδήποτε εσφαλμένη απάντησή μας θα μπορούσε να αμφισβητηθεί ενώπιον του Δικαστήριου της Ένωσης. Μία υπόθεση είναι ήδη στο Δικαστήριο. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι εγκρίνουμε μπορεί να αντέξει το, ε, τον έλεγχο του Δικαστηρίου, διότι ξέρετε ότι είναι πολύ ευαίσθητα θέματα αυτά για τους διοργανωτές που έχουν ισχυρές θέσεις. Αυτά είναι παραδείγματα πρωτοβουλειών, παραδείγματα πρωτοβουλειών που απορρίφθηκαν αλλά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της, της ε, πρωτοβουλίας. Άνεφορο βασικό εισόδημα, Ευρώπη αλληλεγγύης, δημιουργία ε, ενός Ταμείου Ανάπτυξης, σταματήστε της ταυρομαχία, μιλάμε κατά της Πυρηνικής Ένωσης, η Ευρώπη της Εσπεράντο, δημοψήφισμα για τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες και δικαιώματα μειονοτήτων. Αυτά είναι κάποιες περιπτώσεις απορρίψεων. Είναι όλες στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε λεπτομερή περιγραφή των λόγων για τους οποίους ε, αποφασίσαμε όπως αποφασίσαμε. Μετά μας, μου τέθηκε η ερώτηση για τους σερβερ. Εγώ θα έλεγα ότι η ιδιώδης λύση, είπα ποια είναι η ιδιώδης λύση για μένα, ε, δεν έχουμε φτάσει όμως μέχρι εκεί, οπότε μέχρι τότε περιμένουμε και αποφασίσαμε να έχουμε προϋπολογισμό για την Γενική Διεύθυνση Digit που θα τρέχει του σερβερ μέχρι τέλους ε, του 2014, της Ιτίας Επιτροπής δηλαδή. Ελπίζουμε να έχουμε βρει τα χρήματα τότε με επανατοποθέτηση μέσα στην υπηρεσία. Το 2015 Ελπίζουμε ότι και το Κοινοβούλιο που είναι μέρος της Δημοσιονομικής Αρχής να μας βοηθήσει να βρούμε μια μόνιμη λύση. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να σας απαντήσω για το αν είναι πιο δημοφιλής η πρωτοβουλία στη μία ή στην άλλη, στην χώρα. Εγώ Βλέπω ότι οι οργανωτές ε, πρωτοβουλειών κάνουν μείγμα και μεγάλες και μικρές χώρες. Διότι στις μεγάλες χώρες είναι εύκολη η πρόσβαση, αλλά ο κίνδυνος είναι άμα δεν υπολογίσει τη μεγάλη χώρα, ε, άμα δεν μετρήσει, δηλαδή, δεν βγάλει τα νούμερα στη μεγάλη χώρα, χάνει τη χώρα. Οπότε στρέφονται και σε μικρομεσαίες χώρες. Για τα γραφεία τώρα. Είναι οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής. Ε, συχνά, πολύ συχνά ε, ταυτίζονται και με τα γραφεία του Κοινοβουλίου. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μία εκπροσώπηση στα κράτη-μέλη. Στη Γερμανία έχουμε δύο περιφερειακά γραφεία στη Βόνη και το Μόναχο, στη Γαλλία και στη Μασαλία, στην Ιταλία και στο Τωρίνο. Μπορεί να είναι γραφεία δηλαδή μικρά γραφεία των ε, κλιμάκια των ε, γραφείων μας. Uh, asking... Ο κύριος Νταφ ρωτούσε άλλα δύο πράγματα. Το πρώτο το απάντησα. για την έρευνα στα βλαστοκύτταρα. Ήταν το δεύτερο. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα. Το τρίτο ήταν ε, οι δοκιμές σε ζώα οι οργανωτές ήθελαν να παροτρύνουν τη χρησιμοποίηση άλλων μορφών έρευνας για να μειωθεί η χρησιμοποίηση ζώων για δοκιμές, για πειράματα. Για τις ερωτήσεις πολλών μελών για τον τρόπο δημιουργίας των υπογραφών. Εγώ δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα εδώ γιατί ε, το λέει η συνθήκη οπότε απλά πρέπει να περιορίσουμε ίσως τις απαιτήσει, μειώνοντας τον αριθμό των προσωπικών δεδομένων και ξεπερνώντας τα προβλήματα και τους περιορισμούς που επιβάλλονται, Φερπίν, το, το είπα αυτό, ε, το, το πρόβλημα που έχουν ορισμένοι πολίτες που δεν κατοικούν στη χώρα της ηθαγένειάς τους να μετάσχουν στις διαδικασίες. Αυτό θα κάνει πιο το πιο σημαντικό. Ο Μάριο Τενέρο είναι ένας πολύ καλός υπάλληλος, έχω δέψει μαζί του, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ήταν εξαιρετικά καλός και γι' αυτό έφυγε βάσει της κινητικότητας, ασχολήθηκε με ένα νέο φάκελο, μια μεγάλη διάθεση στη Γενική Γραμματεία με στόχο που είχε στόχο να αλλάξει το σύστημα ούτως ώστε κάποιος να είναι υπεύθυνος για ένα φάκελο μέχρι τέλους. Δηλαδή ο στόχος είναι η ίδια ομάδα να εξετάζει το φάκελο από την αρχή μέχρι το τέλος του. Αυτό έγινε πρόσφατα στη Γενική Γραμματεία. Τέλος πάντων, γι' αυτό έφυγε ο Μάριο. Πάντως, οι πρωτοβουλίες είναι ήδη στις γενικές διευθύνσεις. Αυτές είναι που θα ετοιμάζουν την ανακοίνωση, τις απαντήσεις, αλλά στην αναθεώρηση θα γίνει ξανά οριζόντιο θέμα η πρωτοβουλία πολιτών. Τελευταίο ερώτημα Πλάνκοβιτς. οι πρωτοβουλίε συνδέονται με τα βασικά θέματα, τις αλλαγές, ε, προσπαθούν να περάσουν κάποιες τροποποιήσεις. Προφανώς ε, συνδέονται έμεσα με τις ευρωεκλογέ, διότι αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε ότι οι πολίτες ότι τα όργανα δεν είναι μακριά από τους πολίτες, ότι δεν υπάρχει μια ατζέντα των Βρυξελών, αλλά έμεσα αντικατοπτρίζει το πώς θα αισθάνονται οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Απάντησα στον πρόεδρο Κασίνη από τις πρώτες. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ. Εξαιρετικά πλούσια η συζήτηση. Αλλά έφτασαν οι δύο αντιπρόεδροι από τις 4.30. Ζητώ συγγνώμη που σας έβαλα να περιμένετε. Θα Πάμε στο επόμενο θέμα που, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό που είναι η αλλαγή η απόψη του για τις αλλαγές στον κανονισμό για τις ε, ε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Ένα ε, ζήτημα στο οποίο δίνω το λόγο στην κυρία Γκουρμάη αμέσω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι οι συντονιστές συμφώνησαν να επεκταθεί το πεδίο της έκθεσής μου για να συμπεριληφθεί η αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τις γραπτές απαντήσεις στον κανονισμό άρθρα 117 και 118. Η επέκταση αυτή του πεδίου της έκθεσης συνδέεται και με σχετικές τροπολογίες και ο κύριος Καζίνη και η Γραμματεία θα επικοινωνήσουν. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τέτοιες ερωτήσεις, είναι θεμελιώδες δικαίωμα, έχει να κάνει με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και θα σεβαστώ απόλυτα το δικαίωμα αυτό στην έκθεσή μου. Όμως, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τις αυξανόμενες καταχρηστικές πρακτικές από κάποια μέλη αυτού του δικαιώματος και δημιουργήθηκαν ε, ε, καταστάσεις δυσάρεστες. Κάποιοι βουλευτές θέλουν να ε, επηρεάζουν τα στατιστικά στοιχεία με παρεμβάσεις. Αυτό είναι διασπάθηση πόρων και προσπαθειών. Το παράρτημα στους κανόνες 117-118 προβλέπει διάφορες διατάξεις για να προλαμβάνονται καταχρηστικές πρακτικές. Ε, είναι καλή βάση, αλλά δεν αρκεί αυτό όμως. Γι' αυτό υπάρχει τώρα μια νέα απόψη ε, από μένα που λαμβάνει υπόψη δύο τινά. Πρώτον, πώς θα ενισχύσουμε τους υφιστάμενους κανόνες, να τους κάνουμε αποτελεσματικότερους. Ποια πρόσθετα κριτήρια και διατάξεις μπορούμε να εφαρμόσουμε. Για να σας δώσω κάποια στοιχεία. Στοιχεία από το 2011 ε, και, και πιο πρόσφατα έχω να δώσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μελών. Ο μέσος αριθμός ερωτήσεων το 2011 ενός βουλευτή ήταν κάτω από τον μέσο αριθμό ερωτήσεων ε, που θέτει ένας εθνικός βουλευτής ε, στο Βέλγιο για παράδειγμα, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία. Ο συνολικός αριθμός γραπτών ερωτήσεων που κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011 ήταν 12.688 μαζί με ερωτήσεις μη παραδεκτές όπως κρίθηκαν ε, από τον πρόεδρο και αποσύρθηκαν από το μέλος. Ε, το 2011 περίπου 91% των μελών, δηλαδή 676 από τους 736, υπέβαλαν μία τουλάχιστον γραπτή ερώτηση. Ο μέσος αριθμός των ερωτήσεων από, από ένα μέλος μόνο είναι 17. Μόνο 27 μέλη υπέβαλαν πάνω από 17 ερωτήσεις εκείνο το έτος. Ε, αυτά πάνω από τον ε, μέσον όρο είναι το 88% του συνολικού αριθμού των ερωτήσεων το 2011. 11.800 στις περίπου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει αυξανόμενη τάση όπου μικρή ομάδα μελών υπέβαλε σχεδόν όλες τις γραπτές ερωτήσεις, οι καημένοι. Με τέτοια, με αυτή την, γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή στο, στον Τώρα θέλω να σας υποβάλω κάποιες ιδέες για λύση. Κάποιες ιδέες είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που ο Αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς ε, ε, το παίρνει σοβαρά αυτό το θέμα και ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου έκανε επίσης ε, προτάσεις. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσω και εσά πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα και είμαι ανοιχτή σε οποιασδήποτε προτάσεις βελτιωτικές. Ένας τομέας είναι οι ερωτήσεις που είναι πιο αντικειμενικές, ζητάνε δηλαδή στοιχεία, ε, πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη βιβλιοθήκη, το Info και η Κομισιόν εύκολα μπορεί να δώσει απάντηση. Η απάντηση μπορεί να είναι διοικητική από τη διοίκηση. Ε, άλλο, ορισμός του λεγόμενου γενικού συμφέροντος. Πώς θα ε, φροντίσουμε ώστε η ερώτηση που κατατίθεται είναι γενικού συμφέροντος και δεν είναι του συμφέροντος μόνο του ατομικού του βουλευτή που την κάνει. Ε, έχουμε γραπτές δηλώσεις ή ε, προτάσεις ψηφίσματος για να αποφύγουμε τις υποερωτήσεις που θα δυσκολέψουν πολύ την απάντηση. Μια λύση λοιπόν που μπαίνει για να προλάβουμε καταχρηστικές πρακτικές είναι η εφαρμογή μέτρου που θα προβλέπει μέγιστο αριθμό ερωτήσεων. Εγώ θεωρώ ότι στη Βουλή των Λόρδων που είχαν παρόμοιο πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και τις ορθές πρακτικές που υπάρχουν. Εκεί λοιπόν έχουν ένα σύστημα όπου ο αριθμός των ε, ερωτήσεων ε, που εισάγονται ηλεκτρονικά είναι περιορισμένος. Τα μέλη όμως που θα έρθουν ε, και θα έχουν φυσική παρουσία για να υποβάλουν ερώτηση δεν υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Αυτός, αυτό το μέτρο μείωσε τον αριθμό των ερωτήσεων και βελτίωσε το διάλογο και όταν πρόκειται για κριτήρια για το παραδεκτό και έχουν απευθεία διάλογο τα μέλη της Βουλής των, του Λόρδων με τη δίκηση. Είναι λοιπόν συγκεκριμένος αριθμός των ερωτήσεων αναβουλευτή που θα υπολογίζεται σε μηνύα ή διμηνία βάση αλλά αυτό φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα αποδοχής. Μπορεί όμως να έχουμε κάτι παρόμοιο γιατί αν λειτουργεί κάτι καλά σε ένα κράτος γιατί να μην λειτουργήσει και εδώ. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Και για το η σχετικά με το άρθρο 116 του κανονισμού για τις ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κάναμε πολλές διαβουλεύσεις και είμαι ευγνώμων προς εσάς ε, κύριε Αντιπρόεδρε και την ομάδα σας που μας βοηθήσατε. Ο κύριος Ντάφ ζήτησε το λόγο για πρώτος. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Στο πήρα. Καλύτερα να ακούσουμε αμέσως. Καλύτερα να ακούσουμε αμέσως ε, τις θέσεις του αντιπρόεδρου και μετά με εσύ μπορεί να μιλήσεις για πιο πλούσια πράγματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Αν μου επιτρέπετε δύο-τρεις φράσεις. Πρώτα απ' όλα περιμένω και εγώ την έκθεση της κυρίας Γκουρμάη και χαίρομαι που έδειξε προθυμία για αυτή την επέκταση του πεδίου εφαρμογή γιατί είναι ένα θέμα σημαντικό. Και η ώρα των ερωτήσεων ναι. και οι κοινοβουλευτικέ ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετίζονται ημέρα με τι δε στενά. Τώρα, κάποιε ερωτήσει για την ώρα των ερωτήσεων. Αξιολογήθηκε η πρακτική της εφαρμογή από την Κομισιόν, θετικά αξιολογήθηκε. Είδαμε αυτό τον εξάμεινο προγραμματισμό, προετοιμάζονται όλα τα θεσμικά όργανα έτσι πολύ καλά για τις συζητήσεις. Επίσης ε, η πρακτική το 2011, δηλαδή ότι έχουμε ένα βασικό θέμα συζήτησης με τους επιτρόπους, ε, στην ερωτήσεων, εγκρίνεται αυτό ένα μήνα πριν από τη διάσκεψη των Προέδρων ε, και μετά ίσως δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα στη συνέχεια, ιδίω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, που δυσκολεύεται να τηρεί το χρονοδιάγραμμα. ενώ οι επίτροποι μπορούσαν να είναι προετοιμασμένοι και να έρχονται. Οπότε αν ε, γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα πιο πολύ, αυτό θα είναι χρήσιμο ιδίω όταν ε, αναλάβει καθήκοντα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η είδος προγραμματική συζήτηση θα, ήταν χρήσιμη και για το μέλλον. Μία υπόδειξη, νομίζω ότι είδαμε και με τον κύριο Ντάφ στην τελευταία ολομέλη, είναι ότι εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να συζητηθεί ή να τεθεί κατεπηγόντως, το καλύτερο θα ήταν η προφορική ερώτηση μετά συζητήσεως το είδαμε και με το μηχανισμό σταθερότητα ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Και όχι να μπαίνει να να ρωτήσουν την τελευταία στιγμή το θέμα αυτό, που είναι πιο ευρία η συζήτηση με περισσότερου του ενό επιτρόπου. Νομίζω ότι οι συζητήσει αυτέ ε, είναι καλέ να τίθενται σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το πώς μπορούμε και τα δύο αυτά εργαλεία να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και στο μέλλον. Επίσης αυτή η ιδέα ε, για το πιλωτικό αυτό σύστημα, να πειραματιστούμε αυτό το πιλωτικό σύστημα, επιλογή δηλαδή ερωτήσεων με πιλωτικό σύστημα, μπορεί να υπάρξει συμπληρωματική ερώτηση από άλλο ευρωβουλευτή. Έτσι πιστεύω θα είναι γεμάτο και το κοινοβούλιο, το ημικύκλιο, θα γίνεται μια ζωντανή συζήτηση από όλους τους συμμετέχοντες, θα είναι πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επίσης σημειώνουμε με θετικά σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί, αυτόματα να γίνονται γραπτές ερωτήσεις, ε, το να μην δηλαδή γίνει δεκτή αυτή η πρόταση τώρα είναι καλό, αλλά τώρα η πλήρη διαγραφή του παραρτήματος 2 φοβούμε μήπω με αυτόν τον τρόπο διαγραφή και το τμήμα του παραρτήματος που αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Είναι ένα από τα θέματα για τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει ε, στο μέλλον ε, να γίνεται συχνότερη χρήση. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, αλλά αν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, χρησιμοποιούνται έτσι πιο επιλεκτικά και με μεγαλύτερη αυστηρότητα, μπορεί να αποφευχθούν καταχρήσεις, να υποβάλλονται τέτοιες ε, ερωτήσεις μόνο και μόνο για λόγους προβολής δημοσιότητας, και εκεί να βλέπουμε και κάποιες ε, βαθμολογήσεις των ε, βουλευτών, πόσες ερωτήσεις έχει υποβάλει ο καθένας λοιπά. Τώρα, η Επιτροπή για κάποιες προφορίες. 12.971 ερωτήσεις. Θα χτυπήσουμε τις 13.000 σύντομα. Αν διαιρέσετε αυτόν τον αριθμό με τους ε, συναδέλφους, θα δείτε ότι είναι εντυπωσιακό ο αριθμός. Στην πρώτη θέση για φέτος 889 προφορικές ε, ερωτήσεις, τρεις ε, κάθε μέρα δηλαδή, υπέβαλε ο συγκεκριμένος ε, βουλευτής και κάποιες είναι ταυτόσιμες, δηλαδή πως έχει κατάσταση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάδε δίνα χύψη ομέγα χώρας. Έχουμε 300 ερωτήσεις τέτοιου είδους. Δεν ξέρω κατά πόσο με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται οι γνώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά σίγουρα δυσκολεύει πάρα πολύ ε, τις διοικήσεις ε, και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν η κατάσταση αυτή, το να διεκπαιρεώσουν δηλαδή όλους αυτούς τους φακέλους, ε, να τους διαχειριστούν. Γεμίζουν τα ε, ηλεκτρονικά μας ταχυδρομεία και τα γραμματοκιβώτιά μας, πραγματικά κατακλυζόμαστε από τέτοιες ερωτήσεις. Αυτό που προτείνει λοιπόν η κυρία Γκουρμάη δηλαδή ποσοτικός περιορισμό στο των γραπτών ερωτήσεων ανά ή αναπολιτική ομάδα, καλύτερο έλεγχο επιλεξιμότητα, ιδίω όταν υπάρχουν ταυτόσιμε ερωτήσει που στέλνονται απλά και μόνο για να αυξηθεί ο αριθμό των ερωτήσεων που υποβάλλει ο λόγο ή για να πάρει καλή, καλά στατιστικά στοιχεία. Είναι θετικέ οι προτάσεις κυρία Γκουρμάη, θα βοηθήσουν ε, και θα βελτιωθεί νομίζω με τον τρόπο αυτό σημαντικά η κατάσταση. Οπότε Αυτά. Νομίζω ότι μου σύντομος. E Τώρα ο κύριος Ντάφ, ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα το ξαναδούμε αφού πρώτα κατατεθούν οι τροπολογίες. Εγώ σίγουρα θα καταθέσω τροπολογίες. Έχω παρακολουθήσει για αρκετό καιρό το θέμα και από πολύ κοντά, πολύ προσεκτικά. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή την ε, μεταρρύθμιση ε, της διαδικασίας των ερωτήσεων θέλουμε να την έχουμε ολοκληρώσει πριν το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής αυτής περίοδου. Συμφωνώ. Συμφωνώ ως προς το ότι πολλές από αυτές τις ιστοσελίδες που υποτίθεται ότι παρακολουθούν τις επιδόσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά βλέπουν μόνο ε, αυτές τις επιδόσεις με ποσοτικά κριτήρια και όχι με ποιοτικά κριτήρια, Πράγματι, έχετε δίκιο ότι παραπλανούν την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη δηλαδή πιστεύει ότι ο όγκος, ο αριθμός των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων αποτελεί και έναν δίκτυ, αξιόπιστο δείκτη του Βελινεκού στο βουλευτή. Έχω επίσης ε, σημειώσει και κάτι ακόμη, ότι δηλαδή ορισμένες ερωτήσεις απαντώνται, μπορούν δηλαδή να απαντηθούν πολύ απλά αν κάποιος μπει ε, στο διαδίκτυο και κάνει έτσι μια αναζήτηση στην πύλη, τη δικτυακή πύλη Ευρώπη, Europa. Άρα, ίσως θα ήταν καλύτερο να φιλτράρουμε καλύτερα, με πιο αυστηρό τρόπο, αυτές τις ε, ερωτήσεις που είναι πάρα πολύ κοινότοπες ε, ή μπανάλ. και δεν έχουν στόχο να αναζητήσουν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν θα πρέπει το Κοινοβούλιο να γνωρίζει ότι θα μπορούσε να βελτιώσει και τις υπηρεσίες, διότι υπάρχουν ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν πάρα πολύ εύκολα και πολύ πιο φθηνά αν κάποιο ανατρέξει τη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου. Όχι μέσω αυτής της πολύπλοκης ε, αυτής της ε, διαδικασίας που απαιτεί και την παρουσία επιτρόπων. Και έτσι εξοικονομούνται και πόροι οικονομικοί. Αυτό είναι σημαντικό και για μας. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά προσβλέπω ε, στην ε, διεκπαιρέωση αυτού του θέματος το συντομότερο δυνατό. Ο κ. Σέφιν, όχι ο κ. Νταφ που έκανε λάθος να το λέω. κοιτάξτε, αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μου φαίνεται ότι η καρδιά του προβλήματος είναι ότι η εξουσία ε, ε, νέχει και ο κίνδυνο της κατάχρησης. Ε, πρέπει να προλαμβάνουμε τα σπεριτές ερωτήσεις. Ε, όμως ένα κοινοβούλιο τόσο μεγάλο όπως το δικό μας σημαίνει ότι περιορίζεται η δυνατότητα κάθε μέλη να κάνει ερωτήσεις. Αν να περιοριστεί κι άλλο... είναι ένα θέμα. Πολλές φορές ισορεύονται ερωτήσεις ε, γιατί κοιτάζουν ε, τους τους ποσοτικούς προσδιορισμούς. Δηλαδή, πολλές φορές ε, οι άνθρωποι παρακολουθούν ή ο κόσμος παρακολουθεί το έργο του Κοινοβουλίου και μέσα από τις ερωτήσεις. Βέβαια, αυτό σωστό είναι να παρακολουθείτε το έργο, ε, λέω και εγώ πως ο Άντριου ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουμε ποιοτικά κριτήρια. Ποιος όμως θα επιχειρήσει κάτι δύσκολο όταν μπορεί να ε, αποδείξει αυτό που θέλει με ένα κριτήριο πολύ πιο απλό. κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το Κοινοβούλιο, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας ε, το εξηγήσω ε, έτσι με πολλά λόγια, είναι σε μια διαδικασία ομοιογενοποίησης. σε σχέση με τα εθνικά κοινοβουλία σε ορισμένε πτυχέ. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι μία από τι κλασικέ λειτουργίε ε, ενό κοινοβουλίου, που είναι η λειτουργία του ελέγχου, δεν είναι και πολύ αναπτυγμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν υπάρχουν τρε, τρεις κλασικές θεμελιώδεις λειτουργίες για το Κοινοβούλιο, δηλαδή εκλογή, νομοθετική και έλεγχος, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, έχουμε πολύ πιο ανεπτυγμένη την νομοθετική δραστηριότητα και σε σχέση με τις επόμενες ευρωεκλογές προτείνουμε και η εκλογική αρμοδιότητά μας να διευρυνθεί, γιατί θέλουμε την εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν να την συνδέσουμε μια άμεση απόφαση των πολιτών στις διαδικασία, στη δικασία της ευρωεκλο, των ευρωεκλογών και θα πρέπει μετά να δούμε και ποιες ε, διαδικασίες, ποιους μηχανισμούς ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόσουμε για το μέλλον. Η έκθεση του Πάολο Ρανζέλ θα την ε, συζητήσουμε αύριο. Ακριβώς αυτό πραγματεύεται κάποιος από τους πιθανούς μηχανισμούς ελέγχου. Συνεπία της πραγματικής πολιτικής προσαρμογής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνθήκη της Λισαβόνας. Μεταξύ των μηχανισμών ελέγχου, στην προηγούμενη πολιτική μου ζωή ήμουν υπεύθυνο για τις σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Ισπανίας. Τότε αλλά και μετά ο πολλαπλασιασμός των γραπτών ερωτήσεων είχε πάρει εκθετικές ε, διαστάσεις. Δηλαδή αν κάποιος τώρα δει τις γραπτές ε, ερωτήσεις που βάλλονται ε, στις αυτά, στα δύο αυτά χρόνια στην Ισπανική κυβέρνηση είναι γύρω στις 20.000. Γιατί, γιατί υπάρχει μια διπλή τάση. Πρώτον, να υπάρξει μια προβολή μια δημοσιότητα στην εκλογική περιφέρεια του εκάστοτε βουλευτή ή του εθνικού ή του ευρωβουλευτή ανάλογα και δεύτερη τάση, ένα είδος ανταγωνισμού ή συναγωνισμού μεταξύ βουλευτών ή ευρωβουλευτών. Γιατί αν όπως μας είπε πράγματι ο αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς, υπάρχει κάποιος ο οποίος υποβάλλει 800 ερωτήσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να χαίρεται με τον εαυτό όταν έχει υποβάλει μόνο 20. Οπότε φτάνει μια στιγμή που τελικά ξεφεύγουν τα πράγματα. Λοιπόν, από τη μια πλευρά είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα και ικανότητα ελέγχου του Κοινοβουλίου με διάφορους μηχανισμούς μεταξύ των οποίων είναι κάθε είδους ερωτήσεις, εδώ μιλάμε για τις γραπτές. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε αυτή η δυναμική να μην ξεφεύγει και ούτε να χρησιμοποιείται για να μπλοκάρει την Κομισιόν. Θα πρέπει να ταποκριθεί σε αυτή τη δυναμική. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι κάποια εποχή η Υπουργεία της Ισπανικής Κυβέρνησης είχαν κατακλειστεί, διότι έπρεπε να απαντήσουν σε χιλιάδες ερωτήσεις, που πολλές φορές ακριβώς λέγανε η επενδύει στο συγκεκριμένο σημείο για πληθυσμούς πάνω από χιλιάδε, ε, ε, κατοίκους, όλη την Ισπανική επικράτη κτλ. κτλ. να από τους μηχανισμούς, νομίζω το είπε ο κ. Ντάφη, είναι η αναζήτηση στο διαδίκτυο. Κάτι άλλο θα ήταν ο Ευρωβουλευτής που πραγματικά ενδιαφέρεται για κάτι περισσότερο από το να υποβάλει απλά και μόνο μια ερώτηση, να μπορεί να απευθυνθεί ε, στο τμήμα, στη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να πάει ενδεχομένω και αυτοπροσώπους εκεί και να βρει τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι αναζητήσει, τα τα στοιχεία αυτά που επιθυμεί. Να πάει στα αρχεία και να βρει τα στοιχεία κτλ. Έτσι σίγουρα θα φρέναρε κάπως ε, αυτή η κατάχρηση των πρωτοβουλειών που δεν φαίνεται να σημαδεύονται από, ή να χαρακτηρίζονται από πραγματικό ενδιαφέρον απόκτηση ε, γνώσεων και ελέγχου κατά συνέπεια, αλλά απλά το να μπουν σε ένα κατάλογο οι βουλευτές, διότι υπήρξε και μια άλλη πρωτοβουλία που δεν τη κύριος Ντάφ και ο κύριος Σέφιν θα θυμούνται καλύτερα από μένα βέβαια, ότι κάποια στιγμή η Μάρκαριτ Θάτσερ ε, απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση για τις απαντήσεις ε, πλήρωναν ε, για να λάβουν δηλαδή τις απαντήσεις οι βουλευτές για τις απαντήσεις σε που είχαν κάνει. Καλά, σίγουρα αυτό έρχεται σε αντίθεση και με την ίδια την πεπτουσία της του κοινοβουλευτικού έλεγχου, αλλά αυτή η πρόταση υπήρχε από την Θάτσερ. Ευχαριστώ. Κύριο Σχέφνερ Δεν είμαι βέβαιος. Αν ήθελε να το ρωτήσει αυτό πραγματικά ο κύριος Γκερέρο. Τέλος πάντων, το, το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων στην Επιτροπή είναι σημαντικό για κάθε βουλευτή. Όπως ωστόσο κάθε σημαντικό δικαίωμα πρέπει να έχουμε και την ευθύνη της σωστής χρήσης του δικαιώματος αυτού και ευχαριστώ τη Ζήτα για την σωστή προετοιμασία της συζήτηση και για τις και, για τη... και ευχαριστώ τον, κύριο Σευκοβίτση για την ε, εικόνα που μας έδωσε στην κατάσταση. Ε, Ε, το γεγονός ότι ε, δεν επιτρέπεται σωστή προετοιμασία δεν είναι δεδομένο, δεν επιτρέπει να κάνουμε σωστή δουλειά και νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να κάνουμε όσες ερωτήσεις χρειάζονται για την κοινοβουλευτική δουλειά αλλά να μην ανοίξουμε τις δυνατότητες για περαιτέρω καταχρήσεις. Το ποιο είναι το νούμερο αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι λάθος πάντως να νομίζει κανείς ότι μπορεί να εκτιμήσεις ποσοτικά τον, τη δουλειά μας. Αυτή η παρανοήση υπάρχει σε όλο τον κόσμο, αλλά για πολιτικούς και τη δουλειά του Κοινοβουλίου ε, η μέτρηση δεν είναι σωστή. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τον κόσμο να το κάνει, απλά να του εξηγήσουμε ότι μερικέ φορές το ανάποδο σημαίνει. Δηλαδή αυτοί που είναι στα γραφεία μας κάνουν ερωτήσει τη μία πίσω από την άλλη και δεν είναι αυτοί που έρχονται στις συζητήσεις και στα αποτελέσματα του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, ναι, να κάνουμε κάτι. Περιμένω να δω τις συγκεκριμένες προτάσεις του εισηγητή, θα το συζητήσουμε. Ε, ένα σχόλιο έχω μόνο για την ιδέα της κάλπης, της ψηφοφορίας. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να το αφήσεις στην τύχη, αλλά αυτό ισχύει, πρέπει να ισχύει για κάποιες. Όχι για όλες τις περιπτώσεις. Ας πούμε, ε, μπορεί να πούμε ότι επιτρέπουμε μισές ερωτήσεις για τις πολιτικές ομάδες, μισές με κλήρο. Αυτό μπορεί να ήταν μια καλύτερη ιδέα. Ευχαριστώ. Ο Μπρόντς και μετά θα έκλεινα τις παρεμβάσεις και θα έδινα στον Αντιπρόεδρο το χρόνο να κάνει μια σύντομη απάντηση. Ο κ. Μπρόντς. Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να είναι αιτήματα αντικειμενικής ενημέρωσης για να ε, τίθενται, όπως ε, είπε και ο κ. Νταφ, μπορεί να ζητούν ερμηνεία, φράσεις, λέξεις σε ένα κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι κατάχρηση αυτή. Είναι απόλυτα θεμητό να αμφισβητεί κανείς τις εικασίες επί των οποίων εδράζονται πολιτικές ή να επιδιώκονται διευκρινήσεις νοημάτων. Ε, για να μην χάνετε χρόνος, ίσως τα μέλη θα έπρεπε να επισυνάπτουν στις ερωτήσεις την αιτιολόγηση για την ερώτηση. Νομίζω ότι αν υπάρχει χρονοτριβή θα είναι δύσκολο να το δικαιολογούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντιπρόεδρος Εύκοβιτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ εκτιμώ το γεγονός ότι θέσατε το θέμα γιατί όλοι πιστεύουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή σας για την εξέβρεση κατάλληλης λύσης. Βέβαια δεν θα είναι εύκολη η εξέβρεση αυτή, γιατί οι τέσσερις ερωτήσεις αναβουλευτή ένα μήνα ετέθη πριν από καιρό και βέβαια αυτό θα είναι το ανώτατο όριο ή θα θεωρήσουν τα αξιότιμα μέλη ότι υποχρεούνται να τις καταθέσουν αν είναι όριο τέσσερις ερωτήσεις. Αυτές θα είναι υποχρεωτικές. Μπορεί δηλαδή να έχουμε 750 επί 3-4, το θα έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, θα κατακλειστούμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό που προτείνατε να βελτιώσουμε το παραδεκτό, να γίνεται κάποιος έλεγχος, μια εξέταση επίπεδο πολιτικών ομάδων ή όπως είπε ο κ. Ε, ε, Μπρόμς, μια εξήγηση, αιτιολόγηση. Γιατί ένας βουλευτής έχει 300 ερωτήσεις για το ίδιο θέμα ε, ή γιατί είναι τόσες πολλές από πολλές χώρες. Αυτά όλα δείχνουν ότι βλέπουμε με διαφορετικό μάτι την ποσότητα των ερωτήσεων γιατί δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα που μετράει στις ερωτήσεις επίσης και έτσι θα μπορέσουμε να θέσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση. Τέλος, αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, γιατί είναι τριμερής ε, διάλογος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αύριο. Ευχαριστώ για την Επιτροπή σας, για την τεράστια δουλειά που κάνατε στο θέμα αυτό, που απεδείχθη ως θέμα πιο δύσκολο από ό,τι νομίζαμε, αλλά ελπίζουμε ότι αύριο θα μπορέσουμε να βρούμε ε, συμβιβαστική λύση και να προχωρήσουμε με το θεσμικό πακέτο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ελπίζω να προλάβουμε πριν διακόψει τι εργασίε του το Κοινοβούλιο, πριν τελειώσει αυτή η θητεία. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να το πιάσουμε το θέμα μετά τις εκλογές, που σημαίνει ότι θα καθυστερήσουμε 3-4 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για όλη τη δουλειά που κάνατε. Ε, σε αυτό το πολύ δύσκολο φάκελο. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε αύριο να μπορέσουμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος ώστε να έχουμε ε, κίνητρο και δυναμική για να ολοκληρώσουμε και τα άλλα πριν από το τέλος αυτής της θητείας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουρμά για να κλείσει και αυτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί Ακούσαμε ενδιαφέροντα σχόλια που αφορούν τις προφορικές ερωτήσεις ε, και τα πολιτικά κόμματα. Άκουσα πολύ καλές προτάσεις. για να βελτιωθεί η έκθεση. Εγώ αυτό ήθελα να γίνει όταν άρχισα. Βεβαίως όλοι δικαιούνται να κάνουν ερώτηση, αλλά το θέμα είναι πώς ρωτάμε. Ιδιαίτερα όταν δεν μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση ε, από τη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου. Ε, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και δεν είναι όλες ε, ίσες ερωτήσεις. Ελπίζω να βρούμε λύση που θα βοηθήσει όλη τη διαδικασία. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και περιμένω συγκεκριμένες τροπολογίες από εσάς και βέβαια θα έχουμε και καλές συμβαστικές τροπολογίες για να γίνει καλή έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους αγαπητούς συντονιστές που με βοήθησαν να βελτιώσω την έκθεση διότι έτσι θα ωφεληθεί και η μελλοντική μας εργασία που ήδη προϊονίζεται πολύ θετικά πράγματα και σήμερα με την παρουσία του Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς που παρέμεινε για να συζητήσουμε ένα σημαντικό θέμα και ελπίζω να παραμείνει να δούμε τι θα γίνει. ελπίζω να πάει καλά και το θέμα με τα πολιτικά κόμματα. 17 Ιανουαρίου, τα μεσάνυχτα, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, δηλαδή να δώσουμε ένα μήνα από τώρα και ανταλλαγή απόψεων στις 20 και 21 Ιανουαρίου, 24, και και θα ψηφίσουμε στις 11 Φεβρουαρίου. Αν δεν υπάρχουν α, ενστάσεις, αποφασίζουμε έτσι. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς, εξ ονόματος όλων και παρακαλώ τους δύο Αντιπροέδρους να έρθουν εδώ στο βήμα για να αρχίσουμε το επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που επιδείξατε για τη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης. Ε, Βέβαια ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τώρα, ως ήθιστε στην Επιτροπή μας, Έχουμε ακρόαση με τους ε, αντιπρόεδρους που είναι υπεύθυνοι για τη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Ιδίως ό,τι αφορά την ΚΟΖΑΚ, δύο συναντήσεις της ΚΟΖΑΚ ε, πραγματοποιήθηκαν. Δύο ε, συνεδριάσει ολομέλειες δηλαδή. Και είχαμε όμως και δύο συναντήσεις αντιπροσωπιών. Το Δουβλίνο ήταν η πρώτη και στο Βίλνιο στη δεύτερη. Δεν έχουμε συζητήσει τι ε, προέκυψε από τις ε, συναντήσεις αυτές. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη στην Επιτροπή μας. Έγινε συζήτηση και για το άρθρο 13 του Συμφώνου Σταθερότητας. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και συνοπτικά τι έγινε και στη συγκεκριμένη αυτή συνεδρίαση, τι έγγραφα συντάχθηκαν τότε. Να δώσω όμως αμέσως το λόγο στους δύο του Πρόεδρου. Δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει, ο κύριος Μαρτίνες. Λοιπόν, κύριε Μαρτίνες, εσείς ε, κυρίως να μας πείτε για την Κόζακ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Βέβαια και ο κύριος Κάρης ήταν εκεί, έτσι δεν είναι. Και... Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Είναι άλλωστε παράδοση να έρθουμε εδώ να σας κάνουμε έναν απολογισμό, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας, να σας ενημερώσουμε, να ε, είμαστε υπόλογοι αν θέλετε απέναντί σας για το τι έχει γίνει αυτόν τον καιρό. Ίσως είναι η πρώτη φορά, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που και οι δύο αντιπρόεδροι που είναι αρμόδια για σχέσης σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια είμαστε μαζί και οι δύο και αυτό είναι ενδεικτικό για το ότι αυτές οι σχέσεις όλο και πιο πολύπλοκες ε, καθίστανται και αυτό εν μέρη βέβαια αιτιολογείται και από το ότι η συνθήκη της Λισαβόνας όλο και περισσότερο εφαρμόζεται. Και από την άλλη πλευρά θέλω βέβαια να τονίσω την εξαίρετη, τον εξαίρετο τέλειο συντονισμό μεταξύ μου και του κυρίου Κάρας. Στο έργο στο, το οποίο μας ανέθεσε και το Προεδρείο, το Κοινοβουλίο. Σίγουρα διευκολύνθηκε πολύ η δουλειά μας και γιατί είχαμε σε κάθε στιγμή τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων, τον κύριο Καζίν, ήταν στην ομάδα μας, συνεργαστήκαμε τέλεια και βέβαια γιατί και σε αυτό το θέμα αλλά και σε άλλα ενδεχομένω, αλλά σε αυτό σίγουρα το Κοινοβούλιο έχει μια ομάδα υπαλλήλων ε, ικανοτάτων αφοσιωμένων με πολύ μεγάλη εμπειρία. Ορισμένοι ασχολούνται εδώ και χρόνια με το θέμα αυτό. Και μας διευκολύνουν τη δουλειά μας ε, με αξιοσημείωτο τρόπο. Πρέπει να πούμε πολύ ξεκάθαρα ότι τους τελευταίους αυτούς μήνες, ε, όπως είπε και ο πρόεδρος Καζίνη, η δραστηριότητα για την οποία θα κάνουμε τώρα τον απολογισμό, ήταν ουσιώδης. Πολλές συναντήσεις είχαμε, πολλή, πολύ προετοιμασία και φορτωμένη μερίσια διάταξη. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέπω εδώ τον συνάδελφο Κάρας ο οποίος θα πει και αυτός τη δική του εμπειρία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 13 της Δημοσιονομικής Συνθήκης. Στη Λευκοσία το ενέκριναν τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, πέρυσι. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για τις εμπειρίες μας στο πλαίσιο της ΚΟΖΑΚ. Στην Ιρλανδική και στη Λιθανική Προεδρία είχαμε τις συνεδριάσεις αυτές, αλλά θα σας μιλήσω λίγο και για τις διακοινοβουλευτικές διασκέψεις στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής. Το πρώτο νομίζω που πρέπει να πούμε είναι, είναι χωρίς να μπω ε, στην τεκμηρίωση που την έχετε και στη διάθεσή σας, είναι ότι στις δύο συνεδρίες της ΚΟΖΑΚ υπήρξε πολύ σημαντική προσέλευση και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι συμμετείχαν ως ειδικοί ομιλητές, δηλαδή όταν έχουμε τη συζήτηση για τους λεγόμενους keynote speakers, τους βασικούς ομιλητές, νομίζω ότι εδώ πρέπει να αναγνωρίσω μια πολύ σημαντική πρόοδο που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Γιατί πράγματι για κάποιο διάστημα, σε αυτές τις ε, συνεδριάσεις φαινόταν να είναι κάπως επιφυλακτικά τα εθνικά κοινοβούλια, άτομα με εμπειρία, άτομα που ήταν γνωστά ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δεν πολύ ήθελαν ε, οι εθνικοί να μπαίνουν και να λένε τις απόψεις τους σε τα πιο σημαντικά στοιχεία της σημερισιάς διάταξης. Τώρα όμως άλλαξα τα πράγματα. Ο φίλος Νταφ που είναι και σήμερα εδώ συμμετείχε, ο Hans Γκέτ Πέτερινγκ, αυτοπροσώπος, η κυρία Στιφλέρ, Περβάνς Μπερές και εγώ υποφαινόμενος. Μίλησα για διάφορα θέματα που ήταν στη μέση διάταξη. Νομίζω ότι όταν κάνουμε τον απολογισμό δεν πρέπει να το ε, παρακάμψουμε αυτό το γεγονός. Ο τέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Πατ Κόξ, που τώρα προεδρεύει τη Ένωση των τέος ε, Ευρωβουλευτών, ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων. Με πρωτοβουλία μάλιστα των ε, Λιθουανών οικοδεσποτών. Και ο κύριος Κόξ μας εξέφρασε τις απόψεις του και εμβάθυνε στα θέματα της εκλογικής διαδικασίας, των ευρωεκλογών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ενώπιση των ευρωεκλογών του Μαΐου. Οι δύο προεδρίες, η Ιρλανδική και συνεχεία η Λιθουανική, κατέβαλαν εξωσημείωτες προσπάθειες να καινοτομήσουν κατά κάποιο τρόπο δηλαδή αυτές τις δράσεις της ΚΟΖΑΚ να τις βγάλουν έτσι από την τελμάτωση στην οποία είχαν ε, περιπέσει, είχαν γίνει μια ρουτίνα ε, τον τελευταίο καιρό και έτσι σε κάθε μια της περιπτώσεις είχαμε μήματα συζήτησης φόρμη σε σχέση με την κοινότητα των πολιτών, παραδείγματο χάρη ένα φόρμ ε, των νεαρών σε ηλικία πολιτών που εκπροσώπησαν διάφορες σημειονότητες στο Δουβλίνο και είχαμε και μία συνεδρίαση και ανεπίσημη, αλλά μάλλον ανεπίσημη μεν, αλλά πολύ σοβαρή κατά τα άλλα, για τις κοινοβουλευτικές πρακτικές σχετίζονται με τον έλεγχο των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Αρχικά θα συζητεί το μόνο το τι γίνεται σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, αλλά τελικά διευρύνθηκε το πεδίο ε, της συζήτησης. και συζητήθηκαν και τρεις-τέσσερις τομείς όπου βασικά ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ε, εκτελείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με την κυρία Μπερές Είχαμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε ένα φόρουμ γυναικών της ΚΟΖΑΚ. Όπου και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε μια τροπολογία για τα συμπεράσματα και το κείμενο των συμπερασμάτων, η οποία έγινε δεκτή. Έδινε έμφαση αυτό το κείμενο συγκεκριμένα στα ότι τα εθνικά πολιτικά κόμματα, ακολουθώντας κατά κάποιο το μονοπάτι των ευρωπαϊκών κομμάτων, να κάνουν μια προσπάθεια για να υπάρχει καλύτερη γυναική εκπροσώπηση στους εκλογικούς καταλόγους και τις εθνικές και βέβαια και για τις προσεχείς ευρωεκλογές. Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική στιγμή που δεν θα το σημειώσετε εσείς εδώ στη Σταγματική Επιτροπή το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τη γραμματεία της, τη γραμματεία της ΚΟΖΑΚ ανακαινίστηκε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς λειτουργεί αυτή η γραμματεία. Ουσιαστικά ε, υποδέχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς παρέχουμε την ηλεκτροτεχνική υποδομή κτλ. Και νομίζω ότι ήταν ικανοποιητικό η κυρία αυτή από τη Βρετανία που για κάποιους μήνες είχε αυτή τη θέση ε, παρετήθηκε το πάντων για προσωπικούς λόγους και αντικαταστάθηκε συνενετικά από μια άλλη κυρία, την κυρία Φρίντα, του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Φριδά, ίσως ε, θέλει να πει ο κύριος Μαρτίνες, δεν ξέρουμε. durante numerosos ε, años. Ε, Σε οποιαδήποτε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε ότι δικαιολογημένα και όχι αρνητικά επειδή υπήρχε κάποια απογοήτευση από τους ε, βουλευτές για το ποια μπορεί να είναι η συμμετοχή τους ε, στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και σε όλες αυτές τις συναντήσεις ακούσαμε τους συναδέλφους μας στα τεχνικά κοινοβούλια ακούσαμε ότι εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν πιο ενεργά, πιο στενά στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και δι' τις νομοθετικές. Βέβαια πρέπει να δούμε αν γι' αυτό υπάρχουν οι λύσεις και δυνατότητες που προσφέρονται από τις υφιστάμενες συνθήκες ή ενδεχομένως αν όχι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο τροποποίηση των συνθήκων για να επιτρέψουμε αυτή τη συμμετοχή. Στο κείμενο του Δουβλίνου περιλαμβάνονται σημαντικά αιτήματα, παραδείγματος χάρη οι εβδομάδες, οι οκτώ εβδομάδες, αυτή η περίοδος για τις ιτολογημένες γνώμες ε, να γίνουν εβδομάδες το δικαίωμα να ζητούν τα εθνικά κοινοβούλια από την Κομισιόν τροποποίηση ή απόσυρση των προτάσεων της κτλ. κτλ στο Βίλνιους, όπου συζητήθηκαν και προσεχείς ευρωεκλογέ, ετέθη με μεγάλη έμφαση και κατ' εμέ, όχι και τόσο ιταλογημένα πάντοτε, ετέθη λοιπόν το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ένωσης. Οι συνάδελφοί μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια έδιναν συνεχώς έμφαση σε κάποια θέματα σαν κάπως να παραγνωρίζουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού. Εάν δεν συμμετέχουν δηλαδή αυτοί πλήρως, δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση στις διαδικασίες μας. Αυτό που μπορώ να πω, νομίζω ότι καταδεικνύει κατελάχιστον την ανάγκη μεγαλύτερης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ε, και μιας καλύτερης ε, γνώσης των Εθνικών Κοινοβουλίων για το τι κάνουμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν το λέω σε καμία περίπτωση επικριτικά προς τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά η κριτική αν θέλετε στρέφεται σε εμάς τους ίδιους, διότι πολλές φορές αυτή η τόσο μεγάλη άγνοια όχι απλά κάποιον από πολλών συναδέλφων από τα εθνικά κοινοβούλια, μας ε, ξενίζει. Φτάνουν μέχρι κάποιοι να πούν ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών, ε, τον, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου είναι μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τι να πω εγώ, εκπλήσω, αλλά το θέμα είναι γιατί ισχύει κάτι τέτοιο. Διότι βλέπουμε ένα έλλειμμα, όχι δημοκρατικό έλλειμμα γνώσης, το οποίο προκαλείται ακριβώς από την άγνοια, από την έλλειψη γνώσης και από την έλλειψη μηχανισμών πληροφόρησης των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Βουλευτών για το τι κάνουμε εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά υποχρεούνται κατ' εμέ τα Εθνικά Κοινοβούλια και βουλευτέ να γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Όπω και να έχει, Είμαστε απογοητευμένοι σε κάποιο βαθμό. Μπορεί να φαίνεται και από τα λόγια μας και παρόλα αυτά. Την ατμόσφαιρα τη βελτιώσαμε, το κλίμα. Και αυτή θα είναι η κατακλίδα της δικής μου τουλάχιστον παρέμβαση σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, δημοσιονομική, κοινωνική κρίση για τη διαχείριση όλων αυτών από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από το Συμβούλιο. Αλλά και ανεπάρκεια των μηχανισμών που έχουν στη διάθεσή τους τα κοινοβούλια για να ελέγχουν τις κυβερνήσεις τους και για να συμμετέχουν στα νέα αυτά μέσα, στους νέους μηχανισμούς της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης, ετέθησαν όλα αυτά τα θέματα με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Εμείς επιμείναμε, επιμείναμε, λέγω, στο γεύμα που είχα πριν από το συνεδρία του Βίλντος. είπαμε ότι είναι πολύ σαφές το όλο σχήμα. Για να μπορεί να ελέγχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κάθε ένα από τα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχει τον αντιπρόσωπό του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί αυτό δεν κάνουμε καλά και αυτό πρέπει να βελτιώσουμε, εμείς ελέγχουμε το Συμβούλιο συνολικά, εσείς όμως όχι, αλλά ο καθένας από εσάς έχει την ευθύνη να ελέγχει την κυβέρνησή του στο Συμβούλιο. Δεν γίνεται όμως αυτό, ή αν γίνεται, γίνεται με κατακαιρματισμένο και διαφοροποιημένο τρόπο. Υπάρχουν σε κάποιες χώρες βουλευτές οι οποίοι σχέσονται όχι απλά ότι ελέγχουν, αλλά και δίνουν εντολές ε, στην κυβέρνησή τους, συγκεκριμένες και ε, αδιαπραγμάτευτες. Οπότε τι λόγο έχει να πηγαίνει και η κυβέρνηση, να είναι μέλο του Συμβουλίου, γιατί μπορεί να στείλουν απλά ένα mail ή μια επιστολή. Τέλο πάντων, έχουμε αυτό το άκρο και φτάνουμε στο άκρο, άκρο κάποιου που ομολογούν ότι ποτέ στην Εθνική του Βουλή ούτε έλεγχο υπάρχει, ούτε καν απάντηση δεν δίνεται από την κυβέρνηση την ε, για το τι κάνει στη συνεδριά του Συμβουλίου. Τέλος πάντων, είναι προφανές από όλα αυτά ότι καταφέραμε αυτή την επιθετικότητα, ε, αν μπορώ να τη χαρακτήσω, που υπήρχε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να την μετριάσουμε σημαντικά. Και το πετύχαμε αυτό πώς να το πω, αλλάζοντας τη δική μας συμπεριφορά. Εμείς για πολύ καιρό πηγαίναμε στην Κόζακ και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό. Υπήρχε ένα, δύο, τρία εθνικά κοινοβούλια που έπαιρναν το λόγο με πολύ επιθετικό τρόπο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο τι αυτό συνεπάγεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιρνε το λόγο και αντιδρούσε στεναρά ε, κατά αυτών που είχαν μιλήσει με τον επιθετικό αυτό τρόπο. Άρα τι γινόταν, μια αντιπαράθεση, μια σύγκρουση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εθνικά κοινοβούλια και τα άλλα κοινοβούλια δεν έπαιρναν το λόγο για να μην ε, κακοχαρακτηρίσουν τους ε, συναδέλφους τους. Υπάρχουν 4-5 εθνικά κοινοβούλια που επιτίθενται κατά το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, τι κάνουμε τότε, σταματάμε, δεν μιλάμε και τι περιμένουμε. Περιμένουμε να γίνει το ότι 3 ή 4 κοινοβούλια παίρνουν το λόγο και έρχονται σε αντιπαράθεση με αυτά τα Εθνικά Κοινοβούλια που επιτέθηκαν σε εμά. Και έτσι αλλάζουν, τα πράγματα. Γιατί μετά εμεί μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε, εμεί συμφωνούμε αυτό που είπε ο Τάδε Οχύψη Ωμέγα και όχι με τον ΑΒΓ. Και δεν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Γιατί γίνεται πια μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων. Και όχι ε, μεταξύ ημών και του Εθνικού και του Ευρω... των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν είναι συστηματική αυτή την παράτηση που απομονώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στους συναδέλφους του, από τα Εθνικά Κοινοβούλια, με τους οποίους μας συνδέουν δεσμοί, όχι μόνο μέσω της κόζα, καλά, και δυνάμει των ίδιων των συνθήκων, που προβλέπουν ότι υπέρχει να υπάρχει αυτός ο συντονισμός για τον οποίο στον οποίο αναφέρομαι. Τέλος, να σας πω ότι δύο φορές το χρόνο η Κόζακ δημοσιεύει μια έκθεση εξαμηνία έκθεση. Δυστυχώς, δεν είναι πολύ γνωστό αυτό. Παρ' όλα αυτά, οι εκθέσεις αυτές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Διότι δείχνουν κάποια θέματα και την ευαισθησία του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γι' αυτό νομίζω ότι τα οι ευρωβουλευτέ θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, να λαμβάνουν και αυτό το έγγραφο, να το μελετούν. Υπήρχαν συμβουλές ή ιδέες ε, από τον συνάδελφο Ντάφη και από τον Πατ Κόξ στην τελευταία συνεδρίαση της Κόζακ που θεωρώ ότι θα ήταν και αυτές σημαντικές για να ευαισθητοποιήσουμε τους ε, ψηφοφόρους εν των προσεχών ευρωπαϊκών. Πριν ολοκληρώσω, να σας δώσω δύο, ε, να πω δύο κουβέντες για τις δικαιοβουλευτικές ε, διασκέψεις για την ΚΕΠΑ και την ΕΠΑ και στο Δουλό και στο Βιλνιούς σημαντικότατη διακοινοβουλευτική συνεργασία στου τομεί αυτού, βέβαια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν λαμβάνει αποφάσει θέματα εξωτερική πολιτική, όμω εγκρίνει προπολογισμού. Και ελέγχει πάνω απ' όλα τις πρωτοβουλίες που φέρουν το λάβαρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον ημών. Λογοδοτούν οι αρμόδιοι, οι αρμόδιες αρχές. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι ήδη έγιναν τρεις δεκνοβουλευτικές διασκέψεις για το θέμα αυτό και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι δεν δημιουργήσαμε μια νέα συνέλευση. Δεν δημιουργήθηκε μια νέα συνέλευση. Κάποιοι θα το ήθελαν, αλλά Πρόκειται για μία ε, διάσκεψη, η οποία λαμβάνει χώρα σε τακτά διαστήματα και κάθε φορά υπάρχουν άλλες αντιπροσωπείες. Αυτή τη φορά πετύχαμε κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια αντιπροσωπεία με διαφορετικό αριθμό από τις εθνικές αντιπροσωπείες μετά από μακρότητες διαπραγματεύσεις ε, πολλών ετών. Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι και διαφορετική η φύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι ένα ε, απέναντι σε 40 40 γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν δύο βουλές, ε, αλλά τέλος πάντων γιατί είμαστε διαφορετικό κοινοβούλιο. Αυτά είχα να σας πω. Και ολοκληρώνοντας επαναλαμβάνω αυτό που είπα, δηλαδή ότι το κλίμα έχει βελτιωθεί, μεν, αλλά είναι αλήθεια ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση και κάποια εθνικά κοινοβούλια διεκδικούν συστηματικά την ύπαρξη, την καθιέρωση μιας βουλής, αν θέλετε ίσως κάτω βουλής, αντίστοιχα, για τα που θα είναι τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό απορρίφθηκε. Έχει απορριφθεί μέχρι στιγμής. Αλλά είναι δυσάρεστο να συνέρχονται ε, συνεχώς με την πρωτοβουλία ε, του ενός ή του άλλου 8, 10, 15 κοινοβούλια ή αντιπροσωπείες κοινοβουλίων για να συζητήσουν, να προβλέπουν τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, διότι με τον τρόπο αυτό είναι γεγονός ότι δημιουργούνται καταστάσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο Και το γεγονό ότι άνθρωποι όπω ο Άντριου Νταφ θα παρακολουθούν και στη συνέχεια αυτά τα θέματα είναι εγγύηση. Για το ότι θα πρετανεύσει η κοινή λογική και θα βελτιωθούν οι μηχανισμοί γνώσης, πληροφόρηση και θα βελτιωθεί και το κλίμα, η ατμόσφαιρα που δεν θα έπρεπε. Αν και έχει βελτιωθεί, να ε, έχει τέτοιες εκφάσεις σαν αυτές που έχουμε βιώσει. 16 Δεκεμβρίου είναι σήμερα κύριε Πρόεδρε. Αν και δεν πιστε... αυτοί που δεν πιστεύουμε ακόμη, ε, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι η γιορτή της Σάντα Αντέλα, ήταν το όνομα ε, της μητέρας μου, άρα δεν το ξεχνάω. Η Αγία Αδέλα λοιπόν ελπίζω να μας εμπνεύσει. Υπάρχουν και ταινίε ε, με το όνομα Αντέλ. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτά είχα να πω. Α, τι άπιστο είσαι. Μια χαρά πιστό σε ακούω εγώ. Τι να σου πω, θα μπορούσα να πω, μιλήσω και για το Δαλάι Λάμα ή το Βούδα. Τέλο πάντων, δεν θα ξεκινήσουμε θεολογικές συζητήσεις τώρα. Θα μιλήσουμε για τις σχέσεις εθνικών κοινοβουλίων και ευρωπαϊκού. Υπάρχει αυτή η καινοτομία, η νέα συνέλευση της οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ενημερωθούμε για αυτό το καινούριο στοιχείο όπως και για την άλλη ε, συνέλευση. Ο κύριος Κάρας θα μας ενημερώσει και για τα δύο θέματα. Ευχαριστώ. Κυρίες μου και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ο συνάδελφος Μαρτίνες είπε ότι Ίσως θα ξαναμιλήσουμε για την ΚΟΣΑΚ ε, στα πλαίσια αυτής της θητείας μετά τις εκλογές. Σύνθως αλλάζει το 50% των βουλευτών. Η προσωποποιημένη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού με βάση τη δραστηριότητα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς, στη σοσιαλιστική διεθνή, στα συνδικάτα, παντού. Συμμετείχε ο κύριος Μαρτίνας και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία αυτή, γιατί δεν άσκησε μόνο την εντολή του, αλλά με νύχια και με δόντια και με μεγάλη πειθό άσκησε τα καθήκοντά του στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας. Ευχαριστούμε για τις επιτυχίες σου και για όλη σου τη δουλειά. να πω κάτι σημαντικό, βασικό. Έχουμε βέβαια διάφορα επίπεδα συνεργασίας με διαφορετικές νομικές βάσεις. Στην ε, Κόσακ ε, είχαμε και κάποια προβλήματα στην κατανόηση των διαφορετικών ρόλων. Σε ό,τι αφορά το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τη δέσμη των δύο μέτρων, των έξι μέτρων, Ευρωπόλ, ε, ΚΕΠΑ, Όλα αυτά αφορούν μοιρασμένες ε, αρμοδιότητες και όχι μόνο συντονισμό. Και υπάρχει μεν βελτιωμένη κατάσταση, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές παρανοήσεις εις ό,τι αφορά τη συνεργασία στην ε, ΚΟΖΑΚ. Γι' αυτό το θέμα του άρθρου 13 για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το 88 για την Europol, το πρωτόκολλο 2 για την ε, επικουρικότητα και τη συνεργασία στην ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο την ενημέρωση, αλλά και την συνειδητή έλλειψη ενημέρωσης στα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Γιατί Πολλές φορές ε, η κατανόηση είναι ότι σε πολλά θέματα φταίει η Ευρώπη και εμείς εργαζόμεθα σε επίπεδο εθνικό. Δύο είναι οι βασικές αρχές μας όταν κάνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Πρώτον, δεν υπάρχει πολιτική απόφαση αν δεν συμφωνήσουν όλα τα κοινοβουλία. Όλα τα, κοινοβουλία. τα κοινοβούλια συμβάλλουν στο δημοκρατικό έλεγχο, στην δημοκρατική νομιμοποίηση, στη δημοκρατική διαφάνεια. Δεύτερη αρχή. Κάθε κοινοβούλιο είναι αρμόδιο στο επίπεδό του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τις ε, ευρωπαϊκές αποφάσεις, τα εθνικά κοινοβούλια είναι υπεύθυνη για τις εθνικές αποφάσεις. Η τρίτη βασική μας αρχή. Η συνεργασία θα πρέπει να είναι πάνω στη βάση της αρχής της συνένεσης. Ε, δεν είμαστε νομοθέτες στη συνεργασία, αλλά δημιουργούμε δημοκρατικό έλεγχο και νομιμοποίηση, διότι προσδίδουμε διαφάνεια στη συνεργασία τέταρτη βασική αρχή. Θα διευκρινίσουμε το, η διαδικασία του ποιος είναι υπεύθυνο αρμόδιος γιατί όταν στην επόμενη θητεία θα έχουμε μία ε, συνέλευση που θα εδράζεται στο κοινοτικό δίκαιο. Γιατί το δίλημα υπάρχει βέβαια ότι λόγω της ε, κοινωνικής κρίσης, οικονομικής, χρηματοπιστωτικής κρίσης, ε, λόγω όλων αυτών των κρίσεων έπρεπε να δράσουμε σε επίπεδο ένωσης, παρόλο που δεν ε, υπήρχε πάντα η βάση και κάθε δράση χωρίς κοινοτική βάση είναι διακυβερνητική δράση και κάθε διακυβερνητική δράση είναι μία ομόφωνη δράση που περιορίζει τα δικαιώματα του, των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν όλοι να δώσουμε απαντήσεις στις κρίσεις που δεν έχουν τη βάση τους στο ενός ...κυριακό επίπεδο πρέπει να δώσουμε απαντήσεις ε, στην ε, Τρόικα, στον ESM κλπ. σε επίπεδο ένωσης και να ορίσουμε και τις αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Προσπαθούμε λοιπόν ε, στα πλαίσια του άρθρου 33 τη διάσκεψη για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Εγώ ήμουν στις συναντήσεις αυτές μαζί με τον συνάδελφο Μαρτίνες. Όσο περισσότερες αρμοδιότητες έχουμε, τόσο λιγότερο η κατανόηση υπάρχει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Την επόμενη διάσκεψη, 20 με 23 Ιανουαρίου, που θα τη φιλοξενήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να κάνουμε συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, την θέματα συντονισμού οικονομικού, δημοσιονομικού, χρηματοπιστωτικού και να τα συνδέσουμε όλα αυτά με το άρθρο 13, διασκέψεις ή συνεδριάσεις για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και να μιλήσουμε λιγότερο για τη μορφή και περισσότερο για την ουσία. Το περιεχόμενο. Βεβαίως τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τον ίδιο στόχο. Έχουμε τους ίδιους στόχους όταν κάνουμε διάλογο και η εκδήλωση αυτή θα την συγκαλέσουμε από κοινού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα δύο αυτά θα τα συνδέσουμε και με την, τις διακυβερνητικές συνεδριάσεις για το, την, στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής, Εσωτερικής Αγοράς, Κοινωνικής Επιτροπής, Επιτροπής Απασχόλησης, ούτως ώστε να έχουμε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Δεύτερο και διακοινοβουλευτικές επιτροπές μέσα σε ένα τρίμερο. Ε, θα προετοιμάσουμε τη διάσκεψη από 20 με 23 Ιανουαρίου και ελπίζομαι ότι εδώ στο Κοινοβούλιο θα αναδείξουμε ένα μοντέλο για τις μελλοντικέ διασκέψεις. Μία θα γίνεται το, την Άνοιξη, η άλλη θα γίνεται το φθινόπωρο. Ε, δημοσιονομικά θέματα, οικονομική, κοινωνική πολιτική ε, για να έχουμε μια συνολική ανασκόπηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τις επιμεριζόμενες αρμοδιότητες και να ενημερώσουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί αλλιώς οι συναντήσεις που θα οργανώνουμε ε, δεν θα ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, γιατί εδώ μιλάμε για το ρόλο των κοινοβουλίων γενικά στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία η ενίσχυση του ρόλου των κοινοβουλίων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι που πρέπει να μας ενώνει. Και αυτό είναι που δημιουργεί την ανάγκη για τη μελλοντική συνέλευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ξεκινούμε τη συζήτηση για τα δύο αυτά θέματα. Ζήτησαν να μιλήσουν ήδη τρεις συνάδελφοι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε και άλλο θέμα να εξετάσουμε στην μέση διάταξη την έκθεση για τρεμέκη. Παρακαλώ να τηρήσετε τα δύο λεπτά. Νταφ. Θα προσπαθήσω. Να ευχαριστήσω τόσο καταρχάς ε, τους δύο αντιπροέδρους γιατί πραγματικά πιστεύουν στην προσπάθεια να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας και των Εθνικών Κοινοβουλίων. να ευχαριστήσω ιδίω το Μιγγέλ Μαρτίνες που κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών απετέλεσε πηγή έμπνευση για το θέμα αυτό. Έξυπνο, γοητευτικό και σκληρό αν χρειάζεται αντιπρόεδρο, όπως πρέπει. Εκτιμώ την ευκαιρία να που, που μου δόθηκε να μιλήσω σαν βασικός ομιλητής ε, στο Βίλνιους και συμφωνώ ότι η ατμόσφαιρα βελτιώνεται. Υπάρχουν ωστόσο πολλά εθνικά κοινοβούλια ακόμα που αμφισβητούν στην ουσία την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύουν ότι ότι αν ενεργοποιηθεί η κίτρινη κάρτα της επικουρικότητας, τούτο αποτελεί θρίαμβο για τα εθνικά κοινοβούλια, ενώ εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι αποτυχία της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικής και νομοθεσίας. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν την τάση να μην καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου του πώς έχουν τα πράγματα ως προς την αρχή της επικουρικότητας και δεν καταλαβαίνω ότι όλα τα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό συνέχεια και σωστά σωστό είναι αυτό που αναφέρθηκε φοβάμαι ότι αυξάνεται το αίτημα για ένα τρίτο νομοθετικό σώμα που δείχνει ότι δεν καταλαβαίνουν πως ε, η δεύτερη βουλή, το δεύτερο νομοθετικό σώμα αυτή τη στιγμή είναι το Συμβούλιο των Υπουργών. Η τάση της Κόζακ να ψηφίζει συμπεράσματα και συνεισφορές είναι επικίνδυνη κίνηση αν είμαι εδώ στο επόμενο κοινοβούλιο, θα αμφισβητήσω, θα θέσω ερωτηματικά για την παρουσία του κοινοβουλίου σε τέτοιες ψηφοφορίες για τα συμπεράσματα που στο τέλος τέλος προς εμάς απευθύνονται. Είναι λίγο παλαβό λοιπόν και σίγουρα ανατρέπει την αρχή της ε, διάκρισης των εξουσιών να απευθύνουμε εμείς παρατηρήσεις σε εμάς. Και σωστά τα λέει ο κύριος Κάρας ότι πρέπει να στρέψουμε τα εθνικά κοινοβούλια στο να είναι πιο ενεργά και πιο συνεκτικά στην ε, παρακολούθηση του πώς οι κυβερνήσεις του, της κάθε χώρας τηρούν τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις τους. Αυτό δεν το επιτυγχάνω, οπότε δεν μπορούν να αμφισβητούν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια νέα συνέλευση στην επόμενη θητεία που θα ε, αναθεωρήσει τις συνθήκες. Πρόοδος λοιπόν, αλλά και πολλή δουλειά ακόμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουρμάρη. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω κι εγώ. Να τιμήσω κι εγώ έναν άνθρωπο που χάθηκε πριν από λίγο και πριν από λίγες μέρες, τον Νέλσον Μαντέλα Τώρα, για την παρουσίαση των δύο αντιπροέδρων. Πέραν της κρίσεως, η εμπλοκή, η και με αυξανόμενη εμπλοκή νομοθετική της Ευρώπης με τα εθνικά επίπεδα προφανώς έχουν ε, επιπτώσει τη συνεργασία μας με το, με το Εθνικά Κοινοβούλιο. Τρεις παρατηρήσεις. Η δημιουργία συγκεκριμένων τομέων ενδιαφέροντος της Εθνικής Συναντήσης με την ΚΟΖΑΚ δείχνει ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια αρχίζουν να χρησιμοποιούν απόλυτα περισσότερο τη δυνατότητα της διακοινοβουλευτικής συνεργασία. Δεύτερη παρατήρηση, η έμφαση στην οικονομική και χρηματοοικονομική διακυβέρνηση μέσω της ειδική διάσκεψης μιας επιτροπής. Αυτή η επιτροπή, η επιτροπή πάντα ζήτησε, τόνιζε την ανάγκη δημοκρατικού ελέγχου ε, από το Κοινοβούλιο τη οικονομική διακυβέρνηση και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων καθώ και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση τη κρίση. Άρα πρόκειται για ένα καλό βήμα. Και τρίτον, χάρηκα που άκουσα για το, την πρωτοβουλία Φόρουμ Γυναικών για να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή γυναικών βουλευτών και μεγαλύτερη ορατότητα και έμφαση στην ισότητα των φύλων. Να τομίσω ότι το ε, στο Βίλνιους είχαμε ε, μια πρώτη τέτοια συνάντηση και επέτρεψε να έχουμε πολλέ δραστηριότητε στο πλαίσιο μιας άλλη κοινοβουλευτική συνέλευσης, ιδίω τη κοινή συνέλευσης ε, Ένωση ΑΚΕ. Ήμουν πρόεδρο του Φόρουμ των Γυναικών τα τελευταία χρόνια, κάτι που έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή δυνατότητα συζητήσεων, άρα παροτρύνω τέτοιε πρωτοβουλίε. Τελειώνω. Η 18 Δεκεμβρίου θα είναι τα 100 χρόνια τη γέννηση του Βίλι Μπραντ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τώρα που έγινε η συμμαχία ε, ο μεγάλος συνασπισμός με 42% των σοσιαλδημοκρατών γυναίκες ε, καιρός λοιπόν ε, να συγχαρούμε την κυβερνητική κυβέρνηση για μια πραγματικά πολύ καλή συμφωνία μεγάλου συνασπισμού. Πολύ ωραία τα λέπατε Ευχαριστούμε κύριε Μπουρμάη. Ο κύριος Χέφνερ. Ευχαριστώ πολύ. για τις δύο εκτενείς ε, ενημερώσεις. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Ότμαρ Κάρας και συνειδητά θα το ξύνω λίγο, θα το πω λίγο υπερβολικά. Αυτό που επιχειρείται τώρα με αυτή την διακοινοβουλευτική ε, για το δημοσιονομικό σύμφωνο ε, πάει να αντιμετωπίσει μια λάθος εξέλιξη. Αυτή δεν πρέπει να την διαιωνίσουμε, θα πρέπει να ξαναμπούμε σε τροχιά. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, πρέπει να κινηθούμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινότητας και δεύτερον πρέπει να έχουμε ε, μια δημοκρατική τροχιά γιατί αν συνεχίσουμε όπως κάνουμε στο τέλος θα έχουμε μία κουρελού από διάφορα θεσμικά όργανα που δεν θα μπορούν να συντονίζονται ερετά και μη ερετά όργανα και πια δεν θα έχουμε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν που είπε ο Ότμαρ ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να ξαναγυρίσουμε στη λήψη σωστών αποφάσεων, δηλαδή μετά από τον υψηλό βαθμό συνθετότητας που αντιμετωπίσαμε κυρίως μετά τις κρίσεις και φτάσαμε σε διάφορα συστήματα αντιμετώπισης της, τώρα μετά από μία πρώτη φάση ε, αμηχανίας περνάμε σε συντονισμένες ενέργειες μεταξύ μας και μαζί με τους πολίτες για να δούμε αυτή την Ευρώπη πώς θα την τοποθετήσουμε σε μία βάση νομική, μια βάση που θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες και ε, θα λειτουργεί με την κοινωτική μέθοδο και θα προβλέπει αρμοδιότητες με ε, δημοκρατικό τρόπο και το κοινοβούλιο θα είναι ένας χώρος λήψης αποφάσεων ε, όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εδώ, όχι αλλού. Θα ήθελα το κοινοβούλιο αυτό να έχει το θάρρος στο τέλος αυτής της θητείας να πει και να διατυπώσει αυτό που ξέρουμε όλοι, γιατί μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε το δικαίωμα ως κοινοβούλιο να ζητήσουμε μια τέτοια ε, συνέλευση και να κάνουμε προτάσεις ε, για νομοθετικές ε, τροποποιήσεις. Και ο Άντριου Νταφ και εγώ και άλλοι συμμετείχαμε και λάβαμε μια σειρά αποφάσεων που εμέσως καθιστούν απαραίτητη αυτή τη συνέλευση. Η κατανομή των εδρών που μεταρρυθμίστηκε, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο, η έκθεση Ashley Fox για την έδρα του Κοινοβουλίου, Όλα αυτά θα γίνουν μέσα από μια συνέλευση. Και αν πάρουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας και τη δουλειά μας, και τώρα, 4,5 χρόνια μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, αν κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, έναν απολογισμό, θα πούμε ότι σε αυτά και σε αυτά τα σημεία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή της συνθήκης και αυτό θα πρέπει να γίνει ε, με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, της κοινωνίας, των πολιτών και οι συζητήσεις θα πρέπει να έχουν στόχο να χρησιμοποιήσουμε την κοινοτική μέθοδο και με τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών και των κοινοβουλίων τους στο μέλλον να οργανώσουμε την ε, δράση μας σε επίπεδο ένωσης. Αλλιώς θα ε, σταματήσουμε σε έναν τοίχο, σε μια κατακαιρματισμένη ένωση που δεν θα έχει νομιμοποιημένα θεσμικά όργανα, που θα αναλαμβάνει ε, αρμοδιότητες που θα υπησέρχονται στην εθνική κυριαρχία, φορολογική πολιτική, μισθολογική πολιτική κλπ. Όλο και περισσότερο λοιπόν θα χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εμείς θέλουμε τώρα να οργανώσουμε μια διαδικασία δημοκρατική και πολιτική. Ο κύριος Λάινεν που μας τιμά με την παρουσία του εδώ σε μια θέση, σε μια επιτροπή την οποία, στην οποία προείδευε με τόσο καλό τρόπο. Ευχαριστώ. Είχα την τιμή να εκπροσωπώ στην Κόζακ την επιτροπή αυτή επί 7-8 χρόνια σίγουρα και το μήνυμα των δύο αντιπροέδρων είναι σαφές νομίζω. Το διάλογο με τους συναδέλφους μας στα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να τον συνεχίσουμε και να τον ενισχύσουμε. Πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο πολλά για την ενημέρωση σχετικά με τον δικό μας ρόλο στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι τέσσερις βασικές αρχές που ανέφερε ο Ότμαρ Κάρας πρέπει να προβληθούν από εμάς, να αναγνωριστούν από όλους. Και επίσης πρέπει να αναζητήσουμε εταίρους που θα συμμερίζονται τις βασικές αυτές αρχές. Παραδοσιακά υπάρχει μια σειρά εθνικών κοινοβουλίων που καταλαβαίνουν ότι υπάρχει όχι μόνο εθνική αλλά και υπερεθνική δημοκρατία. Το Ιταλικό Κοινοβούλιο το γερμανικό Bundestag, το βελγικό, το αυστριακό κοινοβούλιο και άλλα κοινοβούλια. Είχαμε κοινοβούλια που ήταν κατά της ύπαρξης ενός άλλου διαφορετικού δημοκρατικού επίπεδου, αλλά θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει και μια μεγάλη πλειοψηφία εθνικών βουλευτών, συναδέλφων μας που το δέχονται το επίπεδο αυτό και δεν αποδέχονται την εξέβρεση χειρότερων λύσεων με μικτές αρμοδιότητες που δεν οδηγούν σε ανάληψη ευθυνών. Πρέπει λοιπόν να πούμε στους συναδέλφους ότι θα πρέπει να προασπίσουν αυτήν την αντίληψη για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και ο κύριος Χέφνερ είπε ότι ίσως θα υπάρξει μια νέα συνέλευση, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τις μάχες που θα δοθούν εκεί. Εκπροσώπησα την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέλευσης και μετά και εκεί, Μιγκέλ, το κλίμα ήταν άσχημο. Κάποιοι είχαν απογοητευτεί, αγανακτήσει, γιατί δεν πήραν αυτά που περίμεναν και αυτή η στενοχώρια ή η αγανάκτηση δεν θα είναι λιγότερη αλλά μεγαλύτερη γιατί τα θέματα που θα συζητήσουμε υπησέρχονται ακόμα περισσότερο σε θέματα εθνικής κυριαρχίας. Καλό θα είναι λοιπόν να υπάρξει μια συνέλευση ε, όπου θα, για την οποία θα προετοιμαστούμε και θα δημιουργήσουμε και συμμαχίες για να έχουμε αυτό τον καταμερισμό εργασίας ε, στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου όπως είπαμε τα Εθνικά Κοινοβούλια ελέγχουν τις εθνικές αποφάσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Ευχαριστώ κύριε Σέφλιν. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τους δύο για την Γενική Επισκόπηση. Μία παρατήρηση. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Μαρτίνες, το έλλειμμα πληροφόρησης που αυξάνει άλλα ελλείμματα. Υπήρχε μια στρατηγική επικοινωνία, αν θυμάμαι καλά, που ετοίμαζε η Επιτροπή πριν από 7-8 χρόνια που δεν προχώρησε πολύ μακριά από ό,τι φαντάζομαι. Και η εικόνα που είχα είναι ότι η κοινή γνώμη παραμερίζεται από το εθνικό πλαίσιο, αγνοώντας το τι γίνεται στις Βρυξέλλες, όχι από το Κοινοβούλιο μόνο, γενικά. Η ερώτησή μου είναι, η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη είναι επαρκής, δεν νομίζω ότι είναι. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία για να ε, έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη. Νομίζω ότι αυτό το έλλειμμα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά και να βρει θέση στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Τι, εγώ τίποτα, να ευχαριστήσω όλους σας ήθελα για τα σχόλια δεν είχε, δεν υπήρξε όπως καταλαβαίνετε κάποιο σχόλιο με τον οποίο να διαφωνώ, αλλά κάποιες έτσι μικρές αποχρώσεις. Με ανησυχεί για παράδειγμα και νομίζω ότι το είπε σωστά ο Λάινεν, με ανησυχεί, θα με ανησυχούσε τι πορεία θα ακολουθούσε μία συνέλευση. Η προηγούμενη συνέλευση ήταν περίπλοκη ως προς την λήψη αποφάσεων. Το να κάνουμε τώρα μία συνέλευση μεταξύ 40 ε, δομών ε, όπου και οι 40 θα συμφωνούν είναι παράλογο. Κατά την άποψή μου θα ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει συνένεση μεταξύ των 40 και αυτό το είπε και ο Γιώ. Θα ήταν πολύ δύσκολο να, να υπήρχε συνενετικό αποτέλεσμα σε μια συνέλευση με επαρκή εμβέλεια. Μη βαυκαλιζόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα σε σημαντικό αριθμό κοινοβουλίων υπάρχουν τομείς και κλάδοι, σημαντικοί κλάδοι που είναι αντίθετοι με το σχέδιο οικοδόμηση της Ευρώπης. Καθόλα θεμητό. Εμείς είμαστε με πάθος υπέρ, αλλά πρέπει να αποδεχθούμε ότι υπάρχει κόσμος που είναι κατά. Με πάθος επίσης, ορισμένοι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν σε κάποια κοινοβούλια οι συνάδελφοι αυτοί έχουν την πλειοψηφία, στην πράξη μέσω της ΚΟΖΑΚ αυτό που κάνουν είναι όχι, επικίνδυνο, δεν μπορούμε να το πούμε επικίνδυνο, αλλά θα μπορούσα να πούμε ότι κάποιοι υπάρχουν που στόχο έχουν την δεδηλωμένο στόχο την καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι σύνεπες με τις σκέψεις τους αυτές να θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο είναι ένα καθόλου αναποτελεσματικό και περιττό όργανο, ένα όργανο που θα έπρεπε να καταστραφεί. Με άτομα ε, με τα οποία έχουν ε, διαφωνίες για το τι ερμοδιότητα πρέπει να έχει, μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά με ανθρώπους που πρέπει πιστεύουν ότι το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να πάψει να υπάρχει, ε, τι συζήτηση να κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη ενημέρωση, Τόσο ώστε ένα σημαντικός αριθμός εθνικών βουλευτών να μην πέσουν σε αυτές τις ε, θέσεις. Ότι το κοινοβούλιο είναι ε, ξεδιάντοπη, διεφθαρμένοι, που πρέπει να τους καταργήσουμε. Αυτό είναι αυτά που λένε κάποιοι συνάδελφοι. Όλο και περισσότεροι, να σας πω την αλήθεια. Διότι εσύ είπες κάτι πολύ σημαντικό. Την εποχή σου θυμίζεις ότι υπήρχε ένα, δύο κοινοβούλια όπου κυριαρχούσαν σαφώς αντιευρωπαϊκές θέσεις. Τώρα δεν είναι ένα-δύο, περισσότερα. Και κάποια από τα κοινοβούλια που ήταν πάντα σε μια φιλοευρωπαϊκή γραμμή ε, Τώρα δεν είναι. Είναι σε μια αντιευρωπαϊκή γραμμή. Και έχουν και καλή παρεούλα με αυτούς που ήταν πάντα αντιευρωπαίοι. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα, για να μην σας βάλω, για να τους βάλω σε δύσκολη θέση, αλλά πλιστάκι στον μπορούσα να σας πω ότι εγώ αισθάνθηκα σε πολύ δύσκολη θέση από θέσεις του δικού μου κοινοβουλίου, του Εθνικού Κοινοβουλίου, που ήταν βαθιά διαφορετικές από αυτές που τόσα χρόνια ξέραμε. Όταν η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στόχος αδιαμφισβήτητος στην Ισπανία, η υπογραφή των συνθήκων ψηφίστηκε ομόφωνα στο Κοινοβούλιο. Ομόφωνα, το πρώτο Εθνικό Κοινοβούλιο που ομόφωνα ε, υπερψήφισε την προσχώρηση από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα δεξιά. Αριστερά, συγγνώμη. Όλοι. Τώρα, ο βασικός μου φόβος είναι ότι θα υπάρξει μια σειρά κοινοβουλίων που κάνουν συνεχείς δράσεις, συναντήσεις, συνεδριάσεις, παραμερίζοντας πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας πω δεν θα έλεγα να συνομωτούν, αλλά τέλος πάντων λειτουργούν περιθωριοποιώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αποφάσεις και θέματα όπου το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, αδιαμφισβήτητα. Τέλος πάντων, όπως σας είπα δεν θα πω πολλά πράγματα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα και ε, χρήσιμα να ακούσω του συναδέλφου τη Επιτροπή σα, ε, Είναι από τι πιο ενδιαφέρουσε του Κοινοβουλίου Επιτροπή σα. και καλό θα ήταν το έργο της επιτροπή αυτή, καλό να γίνεται όλο και πιο γνωστό και σεβαστό. Πάντω, να σα πω και κάτι ακόμα. Πρέπει να, να εξετάσουμε τη λειτουργία των, ε, της ΚΟΖΑΚ, του Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα ήμουν τρει ώρε στην Ολομέλεια με τον ε, Ντράγκη. Ούτε 25 δεν ήτανε βουλευτές. Μιλούσε ο Ντράγκη για ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα της ευρωπαϊκής οικονομίας και ούτε 25 δεν ήμασταν. Αφού σκεφτόμουν, είχε η Οικονομική Επιτροπή συνάντηση την ίδια στιγμή. Λοιπόν, ή θα αλλάξουμε τους μηχανισμούς λειτουργίας του Κοινοβουλίου ή απαξιωνόμαστε με τέτοιες συμπεριφορές. Ή το λέμε δημοσία ή σιωπούμε βιώντας μια κατάσταση ανυπόφορη. Συνάδελφοι σύντροφοι, προχωράμε να δούμε πώς θα βγούμε από εδώ πέρα. Ευχαριστώ τον, τον Καζίνη. Κλειδονόμος του Γιολάινεν είσαι και εσύ Παύλο, μην ανησυχείς. Ευχαριστώ. Μα τι λες, εμείς ευχαριστούμε Μιχελάνκελ. Όλοι πλέον είμαστε μάρτινες, μάρτυρες με τη, του, της με το οποία χρωματίζεις τις συναντήσεις. Θα κάνουμε 5 λεπτά διακοπή και μετά την επόμενη συνεχίζουμε με την επόμενη με το επόμενο θέμα στη μέση διάταξη. Rapporto για Έκθεση για Τερμέκη Για τον κανονισμό, για την ανάκληση των, ε, της κοινοβουλευτικής ασυλίας και την άρση. Να, δεν έχουμε πολύ χρόνο. 15 τροπολογίες λάβαμε από την εισηγήτρια από την ίδια τον κύριο Βίλαν και την κυρία Γκαργκάνη. Η κυρία έχει το λόγο. Πρώτο πρώτο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ σύντομη. That, uh, I can support Δεν μπορώ να σας πω ότι στηρίζω όλες τις τροπολογίες πλην τις 17 και τις 18. Γιατί 18 αν γίνει δεκτή θα μας φέρει πίσω στο, στην υφιστάμενη κατάσταση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω. Και μετά για την τροπολογία 17... Ούτε και αυτή θεωρώ ότι είναι καλή. Όλες οι άλλες όμως είναι καλές. Πρέπει να σας πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ασυλία δεν είναι δική μας προνομία, είναι εγγύηση της ανεξαρτησίας και της ακαιρεότητας του Κοινοβουλίου συνολικά. Ένα άλλο θέμα. Η αρμόδια καθήλα Καθήλαρμο επιτροπή, επιτροπή νομικών θεμάτων, εκπροσωπείται εδώ από τον Προεδρό τη. Νομίζω ότι είχαμε καλή συνεργασία, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει το λόγο κάποιος? Λάινεν και μετά Σούλτς. Είμαι σκιώδης για την ομάδα μου, για το θέμα της ασυλίας, σημαντικό θέμα. Στα, στα γρήγορα, συμφωνώ με την κυρία Γιατεμέκη, 17 και 18 να απορριφθούν, γιατί <clears throat> είναι κατά της πρακτικής της Επιτροπής Γιούρη και να δεχτούμε την 21 που είναι λογική συνέπεια. Παράλληλα με τη 17 έχουμε και την τροπολογία 2, είναι η ίδια διατύπωση. 2, 17, 18, όχι λοιπόν, αρνητικό πρόσημο ε, και την 7, γιατί και εκεί είναι μια διατύπωση που δεν είναι καλή. Λέει η απόφαση αυτή για τις αρχές του θυγωμένου κράτους μέλους δεν είναι δεσμευτική. Καλή όμως τις αρχές να συναγάγουν τα ανάλογα συμπεράσματα. Αυτά δεν μπορούν να γραφτούν σε κανονισμό ούτε σε νομικό κείμενο. Είναι πολύ κρυπτογρα... κρυ... απο... αποκρυφικά. Τα υπόλοιπα όμως τα δεχόμαστε. Onorevole Scholz. Scusate, eh, bravo, io sbaglio sempre όχι, όλο λάθος κάνω, συγγνώμη. Εκτός μικροφώνου σχόλιο. Κύριε Μπρόντς, η εισηγήτρια παραπέμπει στο πρωτόκολλο 7 για τα προνόμια και συλλήσεις του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιες, κάποιες ασάφειες. Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι η ασυλία δεν μπορεί να ε, τύχη επίκλησης όταν υπάρχει ε, αυτόφορο αδίκημα, αυτόφωνη πράξη. Και όταν το, έχει το δικαίωμα, το κοινοβούλιο, το δικαίωμα να άρει την ασυλία. Το δεύτερο τμήμα αφορά μόνο την περίπτωση του αυτόφορου και σημαίνει ότι το, το κοινοβούλιο έχει δικαίωμα, καθαρό δικαίωμα άσης η έννοια του αυτοφόρου είναι σαφής όταν μιλάς για φόνο ή κλοπή. Αλλά σε περιπτώσεις αυτό που ο θα χαρακτήριζε ως έγκλημα σκέψης, το αν είναι αυτόφορο ή όχι αμφισβητείται. Αν δείτε το άρθρο 8, αναφέρει ότι οι βουλευτές δεν υπόκεινται σε δίωξη για την άποψη που εκφράζουν, για τι απόψει που εκφράζουν και την άσκηση των καθηκόντων του. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια στην Ολομέλεια, οι φράσει στην Ολομέλεια ή στην Επιτροπή μας τώρα έχουν απόλυτο προνόμιο. Αν εκφράζονται εκτός του Κοινοβουλίου για θέματα αρμοδιότητας της Ένωσης ή ε, όταν η Ένωση κοινοβουλιου για θεματα αρμοδιότητα της ενωσης η οταν η ενωση επιδιωκει μια τέτοια αρμοδιότητα, προφανώς ο Ευρωβουλευτής μιλά ε, ασκώντας τα καθήκοντά του. Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία θα υποβάλω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαργάνη. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της νομικής, αλλά είμαι και αναπληρωματικό μέλος. Να, σχολεί, να συγχαρώ καταρχάς να ευχαριστήσω μάλλον την εισηγήτρια γιατί δέχθηκε τις ε, τροπολογίες της νομικής επιτροπής. Δεν έχω το κείμενο που των τροπολογιών, δεν μου το έδωσε η γραμματεία. Αλλά είπε ότι 17-18 δεν τα δέχεται. Τι είναι για να σχολιάσω αυτό που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. η αλλαγή του κανονισμού και ο στόχος αυτής της αλλαγής είναι να βρούμε στη νομική επιτροπή μια μορφή ενιαίας ερμηνείας του πώς αντιδρούμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις, ούτως ώστε να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ των αντιλήψεων για την ε, άρση της ασυλίας βουλευτών σε εθνικό επίπεδο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Φερρυπίν, οι δηλώσεις ε, βουλευτών. Τι σημαίνει ακριβώς άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή εκτός ε, του βουλευτικού βήματος ένας βουλευτής, ένας ευρωβουλευτής ιδίω σήμερα, έχει ευρείες αρμοδιότητες που εξηγούνται και ασκούνται και εκτός Βρυξελών και Στρασβούργου. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια ισορροπία που θα επιτρέπει μια ενιαία ερμηνεία των ε, καθηκόντων του Κοινοβουλίου. Για το 17 και 18 δεν ξέρω τι είναι, το επαναλαμβάνω, δικές σας τροπολογίες είναι, αν μου πείτε ποιες είναι, η, 17 είναι μια τροπολογία του Σπερώνη. Η 18 είναι μια τροπολογία που έχει και την υπογραφή Γκαργκάνη. Λέει: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνεται είτε επιλογή για κατόπιν ετήσου του διαφορεμένου να εξετάσει σε κάθε στάδιο τη διαδικασία σε μια ληφθήσα απόφαση για άση τη ελευθερία ή για υπεράσπιση τη, αν οι συνθήκε που οδήγησαν στη λήψη τη απόφαση έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά ή αν αυτό δικαιολογείται από τη μέχρι τούδε εξέλιξη τη διαδικασία. Αυτό ήθελα να πω. Αν υπάρχουν νέα στοιχεία, εμείς εξετάζουμε περίπτωση ενό βουλευτή για ένα γεγονός ε, συγκεκριμένο και μετά ο, βουλευτή, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μα έστειλε νέα στοιχεία. Ε, αν δεν έχουν νέα στοιχεία, αν υπάρχει νέο στοιχείο, αν υπάρχει ένα νέο εργαλείο, ένα νέο γεγονός που χρησιμοποιείται κατά, ε, κα, καταχρηστικά, το αγνοούμε. Αλλά θα σε περιπτώσεις νέας δυνατό, νέων στοιχείων θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν αυτή την τροπολογία να τη δεχτείτε, γιατί όταν υπάρχουν νέα στοιχεία, αυτό φοβόμουν ότι αυτό ήταν, γι' αυτό δεν θυμόμουν το νούμερο, αλλά αυτή την εικόνα είχα. Απευθύνω λοιπόν έκκληση να ζητήσω, αν είναι δυνατό, μια ουδέτερη διάφανη διαδικασία ε, ενώπιον ενός νέου γεγονότος που δεν αξιολογείται, που δεν έχει αξιολογηθεί, θα σκόπιμουν η νομική επιτροπή να επανεξετάζει το γεγονός αυτό και να παρουσιάζει την άποψή του. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Τελείωσε ο χρόνος. Χέφνερ, Χέφνερ, τι θέλετε. Ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατος, παρόλο που ζήτησα έγκαιρα το λόγο. Ε, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Γετεμάκη. Σπάνια μπορούμε να συμφωνήσουμε 100% με την άποψη της εισηγήτριας ή διευκρινήσεις και για τη διαδικασία και τους ορισμούς, προθεσμίες κλπ. Όλα είναι σωστά και καλά. Η παρέμβαση του κυρίου Γκαργκάνη εμέσως ε, διευκρινίζει τις διαφορετικές απόψεις και παραδόσεις ε, του δικαίου περί ασυλιών στην Ευρώπη και γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην άσκηση της εντολής στο γερμανικό Bundestag και ήμουν μέλος επί 10 χρόνια της Επιτροπής Ασυλιών. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια πάντα κάναμε άρση της ασυλίας γιατί θεωρούσαμε ότι η ασυλία δεν προστατεύει από ποινικέ διώξεις η ασυλία κανένα βουλευτή και πρέπει να έχει το δικαίωμα να πάει στο δικαστήριο και να αποδείξει την αθωότητά του ο βουλευτής. Ε, και το κοινοβούλιο ε, συνολικά δεν ένιωσε ότι απειλείται. Οπότε πάντα προχωρούσε στην άρση. Υπήρχαν κράτη-μέλη ε, που θεωρούν ότι έχουν ασυλία όταν κατέχουν ένα αξίωμα και κρέμονται από το αξίωμα αυτό θεωρώντας ότι μόνο όταν ε, δεν ε, έχουν το αξίωμα αυτό μπορεί να υπάρξει δίωξη. Εγώ νομίζω ότι η προσέγγιση της έκθεσης είναι πολύ σημαντική γιατί εδράζεται στην πρακτική της νομικής επιτροπής η οποία αποδείχθηκε καλή. Και γι' αυτό η πρόταση είναι πολύ καλή. Τέλος, δύο προσωπικές παρατηρήσεις. Νομίζω ότι το δίκαιο περί ασυλιών ε, προέρχεται από τον 18ο ε, και 19ο αιώνα. Δηλαδή δεν είναι τόσο απαραίτητο σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Γι' αυτό βλέπω με κάποια ανησυχία ότι το γεγονός ότι έχουμε επεκτείνει αυτή την ιδέα της ασυλίας για να περιλάβει όχι μόνο βουλευτές αλλά συχνά και τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους κάθε ε, θεσμικού οργάνου που ξαφνικά απολάβουν ασυλία στα πλαίσια του αξιώματός τους και έτσι δημιουργούνται αμφισβητήσιμες σχέσεις σε σχέση με ε, την αντιμετώπιση ε, μεμονωμένων πράξεων. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, ούτε είναι καλό ότι σε πολλές ε, ε, διεθνικές και πολυεθνικές συμβάσεις η ασυλία ξεπερνά το προσωπικό των πρεσβειών, το αποσπασμένο προσωπικό απεσταλμένο σε μια άλλη χώρα και περιλαμβάνει και άλλες δυνάμεις, ε, ενόπλες δυνάμεις κλπ. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη δηλαδή ε, που πρέπει να την περιορίσουμε. Αυτό ήθελα να πω γιατί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπω ότι ε, υπάρχει αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη. Δύο-τρία λεπτά ακόμα ζητώ υπομονή από τους διασμηνείς, η Να τονίσω ότι η αντίληψη για την ασυλία ποικίλει από κράτος σε κράτος. Η έκθεση δεν αλλάζει την κατάσταση και την κουλτούρα. member states for example if there are criminal cases you are in car accident